Καλημέρα. Χρησιμοποιήστε παρακαλώ τα ακουστικά σας γιατί θα μιλήσω τσεχικά. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας στη συνεδρίαση αυτή της Επιτροπής μας, ε, Υποπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας. Ε, χαιρετώ το προσωπικό, την γραμματεία και βεβαίως τους διερμηνείς μας, λέει ο Πρόεδρος. Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Θα έχετε πάρει την ημερήσια διάταξη φαντάζομαι, οπότε σας ρωτάω κατά πόσο έχει κανείς αντίρρηση στην έγκριση της ημερήσιας διάταξης αυτής. Δεν βλέπω. Συνεπώ, εγκρίνεται. Στη συνέχεια. Πρέπει να εγκρίνουμε τα πρακτικά. Της 25ης και 26ης Ιανουαρίου του 2017. Αν δεν έχετε παρατηρήσεις, θεωρούνται εγκεκριμένα. Και έτσι περνάμε ευθύ αμέσω στο πιο πρώτο θέμα ουσίας που έχουμε σήμερα στην ημερήσια διάταξη, η οποία περιλαμβάνει πολλά. Και το σημείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι θα μιλήσουμε για την αντιμετώπιση των ε, προκλήσεων ασφάλειας που αντιμετωπίζουμε. Εξετάζουμε, για παράδειγμα, τη συνεργασία των ε, ιδιωτικών εταιριών ασφάλειας με τις τακτικές στρατιωτικές μονάδες. Οπότε χαίρομαι πολύ που θα δώσω το λόγο στην κυρία Βάτμαν, την οποία καλωσορίζω εδώ, και θα τη ζητήσω να μας παρουσιάσει όλα τα στοιχεία της ε, εκθεσής σας. Ελάτε εδώ καλύτερα. Δεν σας βλέπω όμως. Πού είσαστε. Α, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ελάτε και σας δίνω το λόγο. Uh, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι πολύ που μου δίνετε ευκαιρία να σας παρουσιάσω σήμερα την έκθεσή μου για τις ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας. Και για να το διευκολύνω αυτό θα χρησιμοποιώ, λέω μελήτρια, τα αρχικά ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας. Yeah. Λοιπόν, ο τομέας αυτός είναι διεθνής. Χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο και απασχολεί πολύ κόσμο. Και φροντίζουν για τη δικιά μας ασφάλεια, όλων μας, τη δικιά σας, τη δικιά μου και όλων μας έχουν πολλέ δραστηριότητες, στρατιωτικέ και μη στρατιωτικέ. και είμαι πεπισμένη ότι στο μέλλον θα παίξουν ακόμα πιο σημαντικό ρόλο, πιο μεγάλο ρόλο. Και υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους πιστεύω ότι η έκθεση αυτή πραγματικά χρειάζεται σήμερα. Πρώτα απ' όλα, Πρόεδρε, το Ευρωβαρόμετρο δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες θέλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Είναι πρώτη τους προτερότητα. Δεύτερον, από την άλλη, βλέπουμε ότι οι επενδύσεις των χωρών μελών δεν φτάνουν στο 2% που έχουμε αποφασίσει για αυτούς τους λόγους. Συνεπώς, οι χώρες μέλη συνεργάζονται όλο και περισσότερο μεταξύ τους για να μειώνεται το κόστος. Σε κάποιε περιπτώσει χρησιμοποιούν λοιπόν οι ιδιωτικέ εταιρείε ασφαλεία οι χώρε μέλη για να πετύχουν ακριβώ το στόχο τη ασφάλεια. Τρίτον, γνωρίζουμε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει ελάχιστη ρύθμιση όσον αφορά την χρήση των ιδιωτικών αυτών εταιρεών ασφαλεία. Επίση, η εκθεσή μου υπογραμμίζει ότι η χρήση των ιδιωτικών αυτών εταιρεών επηρεάζει θετικά ή αρνητικά την εικόνα της Ευρώπης. Οι ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας παίζουν ένα σημαντικό ρόλο προκειμένου να βοηθήσουν τις στρατιωτικές και μη στρατιωτικές υπηρεσίες των χωρών μελών γιατί καλύπτουν το χάσμα που συχνά υπάρχει όσον αφορά το δυναμικό και τις ικανότητες ή επειδή δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα, επειδή ίσως χρειάζονται μερικές φορές και περισσότερες δυνάμεις. Και σε σύγκριση με τις εθνικές ε, δυνάμεις, ιδιωτικές εταιρείες μπορούν να μας βοηθήσουν να εξοικονομήσουμε κόστος, γιατί γνωρίζουν καλύτερα και τι συμβαίνει επί τόπου. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο τέτοιοι ε, φύλακες από ιδιωτικές εταιρείες απασχολούνται από 40.000 ιδιωτικές εταιρείες. Αυτά στην Ευρώπη του 2013. Τα στοιχεία αυτά όμω, τα νούμερα αυτά, μεγαλώνουν όσο περνάει ο χρόνο, λαμβάνοντα υπόψη λοιπόν όλα αυτά τα επιχειρήματα, προφανώ χρειάζεται ρύθμιση, ένα νομικό πλαίσιο και πολιτική ε, υφή αποφάσει. Αρχίζω την έκθεσή μου, ζητάω από την Επιτροπή και από το Συμβούλιο να μα παρουσιάσουν μια επισκόπηση του πού, πότε και για ποιο λόγο έχουν χρησιμοποιηθεί τέτοιε ιδιωτικέ εταιρείε ασφάλεια για να στηρίξουν ευρωπαϊκέ αποστολέ και ζητάμε από τις χώρες μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να μας δώσουν περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την χρήση των εταιριών αυτών προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε μια σωστή αξιολόγηση της χρήσης τους. Τα στοιχεία αυτά θα μας βοηθήσουν στη συνέχεια να αποφασίσουμε πού και πότε η συνεργασία αυτή με τις ιδιωτικές εταιρείες μας εξυπηρετεί είτε οικονομικά, είτε τεχνικά, είτε πολιτικά. Ζητούμε λοιπόν από την Επιτροπή και από το Συμβούλιο να συνεργαστούν με τον ιδιωτικό τομέα στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Για παράδειγμα, ένα σύστημα αναγνώρισης πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να στηρίζει όλες τις χώρες μέλη. Ένα τέτοιο σύστημα θα βοηθούσε την ανταλλαγή πληροφοριών και συνεπώς την ασφαλειά μας άλλα παράδειγμα, με κοινή έρευνα και ανάπτυξη, μπορούμε να προχωρήσουμε και σε κανόνες για την αναγνώριση προσώπων με αυτόματους ελέγχους στα αεροδρόμια, στα μετρό, αλλά και σε άλλα σημεία που συγκεντρώνεται πολλοί κόσμος. Εάν υπάρχουν τα εργαλεία αυτά, στα, αν υπήρχαν στο αεροδρόμιο των Βρυξελών πριν από ένα σχεδόν χρόνο, τότε θα είχαμε γλιτώσει από πολύ πόνο. Οι κάμερες που χρησιμοποιήθηκαν στο αεροδρόμιο δεν μπόρεσαν να δώσουν ε, καθαρή απεικόνηση του τι συνέβη εκεί. Η εικόνα δηλαδή ήταν εθολή. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν όμως τέτοια εργαλεία σωστά, ακόμα και σε πλοία, σε κτίρια. Χρειάζεται φυσικά εκπαίδευση των ε, κατάλληλων δυνάμεων. Συνεπώς, συστήνουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει σε μία πράσινη βίβλο με στόχο την διασφάλιση της συμμετοχής όλων των διαφερομένων μερών από τους δημόσιους και τους ιδιωτικούς τομείς ασφάλειας σε μια ευρεία διαβούλευση. Αυτό θα βοηθούσε προκειμένου να εντοπίσουμε καλύτερα ευκαιρίες για άμεση συνεργασία και προκειμένου να θεσπιστούν οι ελάχιστοι κανόνες δέσμευσης και βέλτιστες πρακτικές. Τέλος, η έκθεση αυτή ζητάει και την ε, δημιουργία προδιαγραφών ποιότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κώδικα και η χρήση των ιδιωτικών εταιριών όμως ε, γίνεται όλο και περισσότερο. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε πάνω σε ένα νομικό πλαίσιο. Συστήνει η εκθεσή μου λοιπόν να ε, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατευθυντήριες γραμμές που να περιγράφουν τις απαιτήσει σε διεθνές επίπεδο αλλά και σε τοπικό επίπεδο που πρέπει να καλύπτουν οι ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας ώστε να μπορούν να υποφεληθούν από συμβόλαιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ζητούμε επίσης από την Επιτροπή να φτιάξει και έναν κατάλογο μια μαύρη λίστα με τις εταιρείε εκείνες οι οποίες δεν έχουν συμμορφωθεί με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Ένα τέτοιο ρυθμιστικό μοντέλο πρέπει βέβαια να διαθέτει ευελιξία. Έτσι, να είναι σαφές αυτό, Πρόεδρε. Σε διεθνές επίπεδο η έκθεση ζητάει από τις χώρες μέλη που δεν το έχουν κάνει μέχρι τώρα να ενταχθούν στο έγγραφο του Μοντρέ όσο γίνεται πιο γρήγορα. Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να συζητηθεί προκειμένου να δημιουργηθεί ένα διεθνές πλαίσιο που θα ρυθμίζει τις δραστηριότητε των ιδιωτικών εταιριών ασφάλειας. Ως εισηγήτρια λοιπόν είμαι υπέρ μιας πιο στενή συνεργασίας μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας. Θα έχουμε πολλές ευκαιρίες, σίγουρα, εάν δημιουργήσουμε ένα νομικό πλαίσιο με διαφάνεια με συγκεκριμένες προδιαγραφές για τον κλάδο και αυτή τη μαύρη λίστα που σας είπα για τους παρόχους οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τις δικές μας προδιαγραφές. Προσβλέπω σε συνεργασία με όλους τους ευρωλευτές μέλη αυτής της Επιτροπής, με τους κοιόδης συζητητές και αναμένω και τις τροπολογίες σας βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε για την πλήρη και διεξοδική αυτή παρουσίαση που κάνατε. Και τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για το ζήτημα αυτό. Θα ήθελα και εγώ να πάρω το λόγο, λέει ο Πρόεδρος, αλλά θα μιλήσω τελευταίος. Ο κύριος Γκάλερ πρώτος, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την συνάδελφο Βάτμαν για αυτό το σχέδιο έκθεσης. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί πρέπει να διεξάγουμε αυτή τη συζήτηση. Sorry, shadow. Όχι, δεν είμαι σκιώδης. Συγγνώμη, συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη. Κοιμάμαι ακόμα, από ό,τι φαίνεται. Με συγχωρείτε. Ναι, λοιπόν, κύριε Γκάλερ, αφού ξεκινήσετε την παρέμβασή σας, να την ολοκληρώσετε. Δεν πειράζει. Ας ξεκινήσουμε πάντως με τους σκιώδεις εισηγητές. Κυρία είναι λοιπόν, είναι η πρώτη. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω λιθουανικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Βάουτμαν, για το σχέδιο έκθεσης που μας παρουσίασε. Πρόκειται για μια εξαιρετική βάση για τις μελλοντικέ συζητήσεις που μπορούμε να κάνουμε για τις ιδιωτικέ εταιρείε ασφάλειας, για την ανάπτυξή τους, για την ανάγκη ρύθμισής τους, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν σύμφωνα με μια μελέτη της Διεθνούς Διαφάνειας όσον αφορά τις ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας και τις ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες που παρουσιάστηκε στην διάσκεψη ασφάλειας του Μονάχου φέτος, οι ιδιωτικές αυτές εταιρείε αναπτύσσονται πάρα πολύ και έχουν περίπου 200 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα. 100.000 περίπου τέτοιες ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας και στρατιωτικές εταιρείες υπάρχουν στον κόσμο και 3,5 εκατομμύρια άτομα απασχολούνται σε εταιρείε αυτέ. Η κυρία Βάτμα μα είπε ότι το 2013 στην Ευρώπη και μόνο είχαμε 1,5 εκατομμύρια προσωπικό σε 40 περίπου χιλιάδες τέτοιες ιδιωτικέ εταιρείες ασφαλείας. Συνήθως έχουμε εξειδικευμένου απόστρατου στι εταιρείε αυτέ, εξειδικευμένου στρατιώτε, επίσης υψηλά ειδικευμένο στρατιωτικό και τεχνικό προσωπικό, έφεδρους στρατιώτες, οι οποίοι απασχολούνται επίσης, οι οποίοι έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν σε στρατιωτικές αποστολές και έχουμε επίσης και στρατιωτικό προσωπικό χαμηλότερης ειδίκευσης. Παγκόσμιες εταιρείες όπως η G4S επεκτείνονται όλο και περισσότερο και θα επεκταθούν ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Ο βασικός λόγος είναι ότι ο αριθμός των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας που για πάρα πολλά χρόνια ήταν βασική αρμοδιότητα των κρατικών ένοπλων δυνάμεων, όλο και μειώνονται. Και οι αρμοδιότητε αυτέ, τα καθήκοντα αυτά, πολλέ φορέ τα εξειδικευμένα αυτά καθήκοντα, καλύπτονται από ιδιωτικέ εταιρείε ασφάλεια. Και ξέρουμε ότι η εξωτερική ανάθεση των αρμοδιοτήτων αυτών χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο, όχι μόνο στι ΗΠΑ, αλλά και στη Γερμανία και σε άλλε χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, μία από τις ε, χώρες αυτές δεν έχει μια συγκεκριμένη ρύθμιση ή ένα σύστημα διοδότησης για τις εταιρείε αυτές, ιδίω όταν αποστέλλονται σε ξένες χώρες, προκειμένου να δραστηριοποιηθούν εκεί. Και έχουμε και συγκεκριμένα παραδείγματα στο Αφγανιστάν, την Αφρική. Συνεπώς, είναι σαφέ ότι χρειάζεται ένα αριθμιστικό πλαίσιο, πρέπει να βελτιωθούν οι κανόνε, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένε απαιτήσει και πρότυπα, τα οποία είναι υποχρεωτικά και δεσμευτικά για όλε αυτέ τι εταιρείε. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που η έκθεση αυτή συντάσσεται από τη δική μα την Επιτροπή και που μπορεί να συζητηθεί από εμά. Βέβαια, ο τρόπο με τον οποίο κάθε χώρα ρυθμίζει τι δραστηριότητε τέτοιων εταιριών σε εσωτερικό επίπεδο αποτελεί εθνική αρμοδιότητα τη κάθε χώρα. Δεν πρέπει όμω να καταλήξουμε σε διαφορετικέ ρυθμίσει για τι χώρε εκείνε, για τι εταιρείε εκείνε οι οποίε δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι εταιρείε αυτέ όταν λειτουργούν σε πλαίσιο υπεργολαβία για συγκεκριμένε χώρε υποδοχή, να δραστηριοποιούνται σε ένα συγκεκριμένο ρυθμιστικό πλαίσιο. Πρέπει λοιπόν να απαντηθούν πολλά ερωτήματα σήμερα. Πρώτον, ποιο είναι ο ρόλο των ιδιωτικών εταιριών ασφάλεια ακριβώ και ποια είναι η νομιμότητα δραστηριοποίησή του και ποιε είναι οι συγκεκριμένε ευθύνε του. Στο παρελθόν, αν ένοπλοι μισθοφόροι από ξένες χώρες συμμετείχαν σε στρατικές επιχειρήσεις σε μία άλλη χώρα και αν αυτοί δεν ε, συμμορφώνονταν με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, πολλές φορές κατάφεραν, κατάφεραν να υπεφεύγουν των ευθυνών τους. Τι γίνεται λοιπόν στις περιπτώσεις εκείνες και πιο συγκεκριμένα ποιες είναι οι ευθύνες των ιδιωτικών εταιριών ασφάλειας που έγκυται ακριβώς η ευθύνη τους και ποια είναι τα όρια των ευθυνών τους αυτών υπάρχει κάποιος, ε, λειτουργούν ως σταθεροποιητικός παράγοντας, πραγματικά συμβάλλουν στην εδραίωση της ειρήνης κάθε φορά που εμπλέκονται σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Και επίσης, θα πρέπει η ρύθμισή τους μάλλον θα πρέπει η ένοπλη αυτή δραστηριότητα να παραμείνει μια εθνική αρμοδιότητα, μπορούν να δραστηριοποιούνται όλο και περισσότερο δυτικέ εταιρείε ασφάλεια. Ξέρετε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε και κάποια παρεμφερή ζητήματα. Θα πρέπει να μειωθεί το μέγεθος των εταιριών αυτών. Ορισμένες από τις εταιρείε αυτές μπορούν να αποτελέσουν μικρούς ειδικευμένους στρατούς, αν δεν περιορίσουμε τελικά το μέγεθός τους. Επίσης, ποιες υπηρεσίες μπορούν να παρέχουν. Αυτή τη στιγμή οι υπηρεσίες τους καλύπτουν ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Τρίτον, Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ε, συμμετοχή των ε, ιδιωτικών εταιριών ασφαλείας και των ιδιωτικών στρατιωτικών εταιριών σε αποστολές των Ηνωμένων Εθνών και σε αποστολές και ΕΠΑ. Όταν παρέχουν ε, οι υπηρεσίες αυτές φρούρησης σε αντιπροσωπείες των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς ακριβώς πρέπει να ρυθμίζεται η δραστηριότητά τους. Συμφωνώ με τις προτάσεις που κάνει η δραστηριότητα προκειμένου να έχουμε κοινέ κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τη δραστηριότητα των εταιριών αυτών. Επίσης στηρίζω την ιδέα ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πράσινη βίβλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να υπάρχουν συγκεκριμένα πρότυπα και πρότυπα ποιότητο για την παροχή των υπηρεσιών αυτών, τουλάχιστον για τον τομέα εκείνο που είχε να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνεται βέβαια και μία πρόταση για τη δημιουργία ενό ε, μαύρου καταλόγου για τι ε, εταιρείε αυτέ, οι οποίε δεν συμμορφώνονται με συγκεκριμένου κανόνε. Πολύ φοβάμαι όμω ότι ο κατάλογο αυτό μπορεί τελικά να είναι αντιπαραγωγικό. Δεν μπορώ πάλι όμως να απορρίψω και την πρόταση αυτή της εισηγήτριας. Επίσης, ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας λειτουργούν τόσο στη θάλασσα όσο και στην επικράτεια των κρατών μελών. Πρέπει λοιπόν εδώ πέρα να δούμε πραγματικά πώς θα ρυθμίσει τη δραστηριότητά τους. Όταν δραστηριοποιούνται στη θάλασσα οι ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας, οι φρουροί αυτοί δεν θα πρέπει να παραμένουν πάνω στο σκάφος γιατί ενδεχομένω να μπορεί να συλληφθούν, ενδεχομένως δεν μπορούν να μπουν στα εθνικά χωρικά, χωρικά ύδατα συγκεκριμένων χωρών. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να εμφανίζονται περισσότερο στην έκθεση αυτή και οι δραστηριότητε στη θάλασσα των ιδιωτικών αυτών εταιριών ασφάλεια. Εκκρεμούν πάρα πολλά ερωτήματα, δεν έχουν δοθεί ακόμα αρκετέ απαντήσει. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε καταρχά ποιο θα πρέπει να είναι το πεδίο εφαρμογή τη έκθεση αυτή. Θέλουμε απλώ συστάσει, θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα δεσμευτικό πλαίσιο. Ποιο είναι ακριβώ το φάσμα των δραστηριοτήτων που θα καλύπτεται από τι ιδιωτικέ αυτέ εταιρείε ασφάλεια. Στο παρελθόν, μην ξεχνάμε, ορισμένε από τι αρμοδιότητε αυτέ πριν από 15-20 χρόνια ήταν αρμοδιότητα μόνο των κρατών μελών, των εθνικών στρατών. Αναφερόμαστε εδώ πέρα σε έναν κλάδο που αναπτύσσεται όλο και περισσότερο, είναι ιδιαίτερα κερδοφόρου. Οι εταιρείε αυτέ αναπτύσσουν όλο και περισσότερο τι δραστηριότητέ του. Πολλέ φορέ ξεφεύγουν από τον εθνικό έλεγχο. Θα πρέπει να περιορίσουμε λοιπόν το μέγεθο των εταιρεών αυτών, θα πρέπει να περιορίσουμε το εύρο των δραστηριοτήτων του, προκειμένου οι εταιρείε αυτέ να μην προκαλέσουν προβλήματα ασφάλεια. Σα ευχαριστώ πολύ κυρία Βάουτμαντ, λοιπόν για το σχέδιο αυτοέκθεση και η δική μου ομάδα, το ΕΛΚ, θα συμμετάσχει ενεργά στην εκπόνηση έκθεση αυτή με την καταβολή, υποβολή με συγχωρείτε τροπολογιών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φανζολίκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, είναι πάρα πολύ σημαντικό μετά τον εισηγητή να δίνετε το λόγο στους κοιόδης Νομίζω ότι είναι ένας καλός κανόνας και ευχαριστώ κύριε Γκάλε που καταλάβατε και κατανοήσατε τη θέση μου και νομίζω ότι εντάξει αφού το είπα μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε με τις παρεμβάσεις μας. Συνάδελφοι, θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς την εισηγήτρια, την κυρία Βάουτμαντς για αυτήν την εξαιρετική προσπάθειά της. Υπάρχουν κάποιες διαστάσεις του θέματος που προσεγγίζει η ε, συγκεκριά με τις οποίες συμφωνώ. Ιδίως όσον αφορά τα, αριθμητικά στοιχεία των εργαζομένων στις ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας που αυξάνονται και λαμβανούμε υπόψη και των διεθνικών επιπτώσεων, την ε, έλλειψη, την απουσία ευρωπαϊκού νομοθετικού πλησίου που δημιουργεί προβλήματα για το περιβάλλον ασφάλειας. Ιδίω αν λάβουμε υπόψη την ανεπαρκή διαφάνεια, παρακολούθηση αλλά και την ε, κλίση σε λογοδοσία αυτών των ιδιωτικών εταιριών ασφάλειας και στρατιωτικών εταιριών. Σε αυτό το πλαίσιο χρειάζεται μια αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης γύρω από αυτές τις ιδιωτικές ε, εταιρείες ασφάλειας που δραστηριοποιούνται ή έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε, τρεις, σε τρίτες χώρες ή προσφέροντας υπηρεσίες τους σε ευρωπαϊκές μονάδες. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι κοινό σκοπός τόσο των θεσμικών οργάνων όσο και των κρατών μελών προκειμένου να διαμορφωθεί μια συνολική εικόνα των δομών που δραστηριοποιούνται στις υπηρεσίες ασφάλειας. Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα είναι ότι η χρήση ιδιωτικών εταιριών ασφαλειών χρειάζεται σε τελική ανάλυση να ε, διέπεται από κοινωνικά και ηθικά χαρακτηριστικά, ιδίως όσον αφορά ε, του, τις αμοιβέ των εργαζομένων τους, αλλά και ε, όσον αφορά εκείνους με τους οποίους έρχονται σε επαφή στι τρίτες χώρες και αναφέρομαι στου πληθυσμού, αλλά και τις αρχές αυτών των κρατών. Αυτό σχετίζεται και με τη, τα νομικά κενά που υπάρχουν όσον αφορά τη δραστηριοποίηση αυτών των ιδιωτικών εταιριών ασφαλεία σε τρίτε χώρε. Επίση, η κοστοαποδοτικότητα δεν πρέπει να είναι το βασικό κριτήριο όσον αφορά τα ζητήματα ασφαλείας μια προσεκτική αξιολόγηση των ε, συστημάτων ιδιωτικοποίησης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τους κινδύνους. Λόγω της ε, μεταβελόμενης δυναμικής γύρω από την ασφάλεια νομίζω ότι ο αποτελεσματικός έλεγχος μέσω της εφαρμογής σαφών και αυστηρών κανόνων για τις ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν μπορούμε να δεχθούμε ευρωπαϊκές εταιρείες να συνδέονται με απάνθρωπες πρακτικές σε τρίτες χώρες. Τέλος, οι ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας δεν προσφέρουν μόνο καθαρά ε, υπηρεσίες ασφάλειας, αλλά πολλές φορές ε, συλλέγουν και πληροφορίες. Και αυτό σημαίνει ότι αναπτύσσουν ικανότητες πληροφόρησης οι οποίες επίσης θα πρέπει να ελέγχονται και να ρυθμίζονται νομοθετικά. Άλλη μια φορά να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και προσβλέπω στη συνεργασία μαζί της, με εκείνη και με όλους τους σκιώδεις εισηγητές για αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Ευχαριστώ κύριε Φραντζόλικα. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Μπούχνερ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Το θέμα είναι τα βασικά δικαιώματα, τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ιδιωτικοποίηση της ασφάλειας και της άμυνας έχει επιφέρει τα τελευταία χρόνια αρνητικότατες επιπτώσεις. Ναι, είναι ακριβό το να πληρώνει κανείς αστυνομικούς και στρατιωτικούς. Αλλά ποια είναι η αξία σε τελική ανάλυση μιας πολιτικής ασφάλειας και άμυνας που θα προέρχεται από και θα πηγάζει από τον ίδιο τον λαό ιστορικά. Πρόκειται για κατάκτηση του δημοκρατικού κράτους δικαίου το να υπάρχει αυτός ο έλεγχος από τα κάτω. Ας μην αυταπατώμαστε. Μια ιδιωτική εταιρεία ασφάλειας μπορεί να παρέχει και καλές υπηρεσίες, αλλά κινητήρια δύναμή της θα είναι πάντοτε η ε, επίτευξη του μέγιστου δυνατού κέρδους και όχι η προστασία των συνταγματικών ε, επιταγών. Κάποιες φορές μπορούν αυτά τα πράγματα να συμβαδίζουν, κάποιες φορές όμως και όχι. Βεβαίω η κατάσταση έχει πάρει μια συγκεκριμένη τροπή. Αλλά πρέπει κοινωνικά να δούμε ποιε επιπτώσεις θα έχει. Υπάρχουν δυστυχώς πολλά μαύρα πρόβατα σε ε, αυτόν τον τομέα. Υπάρχει η εμπειρία της Blackboard στο Ιράκ. Υπάρχουν οι εγκληματικές πράξεις ε, ανθρώπων ε, που έχουν ε, αποκαλυφθεί τα τελευταία χρόνια. Και εδώ στη Δυτική Ευρώπη, άνθρωποι που προέρχονται από τη Δυτική Ευρώπη. Και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχαμε αρνητικές εμπειρίες, αρνητική πείρα με ιδιωτική εταιρεία ασφάλειας. Ήταν φτηνή, ήταν φτηνή και ως προς τις αμοιβέ που παρέχει στους εργαζόμενους και τι συνέβη, τρεις ένοπλες επιθέσεις είχαμε εκείνη την περίοδο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάποιοι δεν θα το ε, θυμούνται, αλλά είχαν κλαπεί κάτω από τα μάτια της ίδιας της αυτής ιδιωτικής εταιρείας ασφάλειας ε, πάρα πολλά έπιπλα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ναι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε πληγεί ως προς τη φήμη του τότε ως δημοκρατικά εκλεγμένο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και με αυτό θα ήθελα να περάσω στις παραγράφους 1 έως 4. Και θέλω να πω ότι η βασική μου κριτική είναι ότι σε αυτές τις ε, παραγράφους το βασικό επιχείρημα είναι η εξοικονόμηση χρημάτων. Όπως είπα και με τα όσα ε, ανέφερα δεν συμφωνώ καθόλου. Δεν είναι δυνατόν, δεν διανοούμε σε αυτόν τον τομέα να γίνεται λόγος για εξοικονόμηση πόρων, διότι η, δυστυχώς οι αρνητικές επιπτώσεις της εξοικονόμησης πόρων και χρημάτων σε αυτόν τον τομέα είναι υπερβολικά ε, μεγάλες. Το ίδιο ισχύει και για τις αιτιολογικές σκέψεις P και Q. Όπως γνωρίζετε, καθώς το έχουμε συζητήσει εδώ στο Κοινοβούλιο, υπάρχουν διπλωματικές συγκρούσεις μεταξύ κρατών μελών της Ένωσης και της Ινδίας, για παράδειγμα. Για το γεγονός ότι ε, η, οποία, η ε, Ινδία ε, συνέλαβε εργαζόμενους ιδιωτικών στρατιωτικών εταιριών που κινούνταν στα χωρικά ύδατά της και υπάρχει κατηγορία ότι αλληλείς της Ινδίας δολοφονήθηκαν από πειρά εργαζομένων τέτοιων ιδιωτικών ε, στρατιωτικών εταιρεών ε, της Ευρώπης. Και ε, είναι γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί εισήλθαν στα χωρικά ύδατα κυριαρχού κράτους. Αυτό το κόστος ποιος θα το εκτιμήσει. Στην αιτιολογική σκέψη Β. Υπάρχει μια σημαντική ε, έννοια. Υπάρχει ε, η, ε, η γνώση πλέον ότι έχουν ιδρυθεί ιδιωτικές στρατιωτικές ασφάλειες, εταιρείες ασφάλειας προκειμένου να μπορέσουν να παρακάμψουν το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει. Επίσης, υποστηρίζω το αίτημα να καταρτιστούν κατευθυντήρες γραμμές της παραγράφου 4 και το αίτημα ε, για την θέσπιση πιστοποιημένων παρόχων υπηρεσιών. Σε ό,τι αφορά την, ε, τις, ε, προδιαγραφές ποιότητας, συμφωνώ επίσης. Χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα ευέλικτο και ασφαλές ρυθμιστικό πλαίσιο. Και αυτό είναι πράγματι ένα από τα κεντρικά σημεία της εισήγηση. Γι' αυτό και πιστεύω ότι πρέπει να γίνουμε ακόμη πιο σαφεί και πιστεύω ότι για το σκοπό αυτό χρειαζόμαστε οδηγία ή κανονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να τονίσουμε ότι ο χρόνος τρέχει, διότι εδώ και χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα, ενώ παράλληλα ο αριθμός των εταιριών αυξάνεται και τελικά διαμορφώνεται ένα σκηνικό άγριας δύσης. Επίσης η παράγραφος 15 αναφέρει κάτι πολύ σημαντικό που θα μπορούσαμε να το δούμε και αποκοινούμε την παράγραφο 18. Το ζήτημα μιας πραγματικά αποτελεσματικής ε, διεθνούς ρύθμισης του θέματος. Και εδώ ο χρόνος έχει ε, περάσει. Χρειάζεται άμεσα μια ε, διεθνής σύμβαση που θα ρυθμίζει τα θέματα αυτά. Αυτά από μένα και σας ε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπίχνερ. Κυρίες και κύριοι. Έχουμε πέντε ακόμα ομιλητές στον κατάλογο, οπότε σας παρακαλώ πολύ όλους να μην μακρηγορείτε. Επόμενος Σκιώδης ο κύριος ε, Σάπσχάουζερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλές παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, συμφωνώ με αυτά που είπε μόλις ο συνάδελφος. Και εγώ πάω προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως, πρώτα απ' όλα να κάνω μια παρατήρηση ουσίας. Έχουμε να κάνουμε με τη σέβαση του Μοντρέ εδώ. Έχουμε να κάνουμε με μια διεθνή συνεργασία που ήδη υπάρχει. Οπότε αναρωτιέμαι γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση και το κοινοβούλιο μας προσπαθεί να προσθέσει κάτι. Έχουμε να κάνουμε με κάτι διεθνές, με διεθνή σύμβαση, οπότε εμείς τι έχουμε να προσφέρουμε παραπάνω. Η Ευρώπη για άλλη μια φορά θέλει να χώνει τη μύτη της παντού. Και γιατί, γιατί υπάρχει ίσως αυτή η ιδέα της Ευρωπαϊκής Άμυνας, αλλά ειλικρινά εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί ανακατευόμαστε σε αυτό το ζήτημα. Τώρα, επί της ουσίας, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια διάκριση που την κάνει και ε, το κείμενο του Μοντρέ. Υπάρχουν ιδιωτικέ εταιρείε ασφάλειας που είναι όπως αυτές που φιλούν μια τράπεζα ή κάτι άλλο, αλλά υπάρχουν και ιδιωτικέ εταιρείε ασφαλεία οι οποίε δραστηριοποιούνται σε εμπόλεμε περιοχέ. Και εδώ περί αυτού πρόκειται. Πρόκειται δηλαδή για ιδιωτικέ εταιρείε ασφάλεια, οι οποίε ε, με κάποιο τρόπο, άμεσα ή έμεσα, δρούν εκ μέρου των χωρών μελών. Εγώ είμαι βασικά κατά τη αρχή αυτή. Είμαι απόλυτα κατά τη αρχή αυτή. Γιατί καταλήγουμε σε μια περίεργη κοινωνία, ακριβώς θέλοντας να κάνουμε εξοικονομήσεις, ιδιωτικοποίησαμε το δίκαιο συμβάσεις εννοώ με τον Καναδά, η ΣΕΤΑ για παράδειγμα, στο όνομα της οικονομίας τώρα θέλουμε να ιδιωτικοποιήσουμε και τις ένοπλες δυνάμεις. Ενώ ένα κράτος δικαίου, δικαίου πρέπει να έχει το μονοπόλιο της ε, εξουσίας αυτής της ένοπλης. Τώρα λοιπόν θα έχουμε ιδιωτικέ εταιρείε που θα παραμβαίνουν και η εθνική κυριαρχία, η δημοκρατία θα κάθονται ανήμποροι και θα κοιτούν κάτι το οποίο τους ξεφεύγει και από πλευράς δικαίου, γιατί θα είναι ιδιωτικό το δίκαιο αυτό σε διεθνές επίπεδο, αλλά και όσον αφορά την ενοπλή παρέμβαση. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε με τίποτα. Ο συνάδελφος πολύ σωστά αναφέρθηκε στις καταχρήσεις, στις Blackwater για παράδειγμα, που άλλαξε όνομα πολλές φορές προκειμένου να χαίρει κάποιας νομιμότητας. Αλλά αυτό που είναι ακόμα πιο σοβαρό πιστεύω είναι η χρήση από τις χώρες μέλη των ιδιωτικών αυτών εταιριών ασφάλειας για να ξεφεύγουν από το δίκαιο. Εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να φτάσουμε στη διάλυση του κράτους μέσω της ασφάλειας, της άμυνας. και όλων όσων έχουν να κάνουν με το μονοπόλιο των χωρών. Αλλιώ δεν θα έχουμε χώρε. Το κράτο δικαίου τελικά θα είναι ένα κράτος χωρί δίκαιο. Εκεί θα καταλήξουμε. Όλα αυτά ήθελα να υπογραμμίσω τώρα για τι παρατηρήσεις. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια αρμοδιότητα που είναι των χωρών μελών. Έχουμε ανακατέψει το διεθνές επίπεδο. Βάζουμε και την Κομισιόν γιατί τα θέλουμε όλα αυτά να τα κάνουμε πιο ηθικά, αλλά τελικά ο τελικός στόχος είναι για άλλη μια φορά να αφαιρέσουμε από τις χώρες μέλη μια αρμοδιότητα λέγοντας ότι η Επιτροπή θα τα βοηθήσει. Τα κάνουμε αυτά αρμοδιότητα της Κομισιόν, λέγοντας ότι για να διευκολύνει τις χώρες μέλη θα αναλάβει μια αποστολή που δεν την έχει τώρα, έτσι, προσοχή. Οι πληροφορίες δεν είναι θέμα ε, κομισιόν είναι θέμα των χωρών μελών. Δεν έχει δικέ της δυνατότητε πληροφοριών η Κομισιόν. Για άλλη μια φορά λοιπόν κάνουμε μια προσπάθεια να διαλύσουμε τις χώρες, να τους αφαιρέσουμε αρμοδιότητες και αυτό αποτελεί τελικά επίθεση κατά της κυριαρχίας των λαών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γκάλερ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ Πολύ σύντομα, συμπληρωματικά προς αυτά που είπε η σκιώδης του ΕΛΚ και συμφωνώ με όλα όσα είπε. Ε, είπε ότι εξακολουθούν να παραμένουν ανοιχτά ορισμένα ερωτήματα. Συμφωνώ και εγώ. Καθήκον μας είναι να δώσουμε απαντήσεις για το ποια θα πρέπει να είναι η πορεία μας από εδώ και μπρος, η κατεύθυνση που θα υιοθετήσουμε. Υπάρχουν βεβαίως και κάποιοι ε, τομείς που δεν αφορούν απαραίτητα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποια ιδιωτική εταιρεία που φυλάσει μια άλλη ε, ε, ιδιωτική εταιρεία δεν χρειάζεται σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος και στο πλαίσιο της ένομης τάξης του δεν χρειάζεται να ε, ρυθμίζεται από κανονισμό ή οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα βεβαίως και από την άλλη πλευρά ε, ισχύει ότι μια ευρωπαϊκή αποστολή δεν μπορεί να φυλάσσεται από ε, μονάδα κράτους μέλους και μόνο. Φυσικά σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται να έχουμε τη δυνατότητα να προσλαμβάνουμε ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας οι οποίες, οι οποίες να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές. Και εκεί πράγματι χρειάζεται ρυθμιστικό πλαίσιο. Αυτό που πρέπει να μας αποσχολήσει είναι σε ποιον βαθμό θα αποφασίσουμε να ε, αναθέσουμε... Ε, αρμοδιότητες που κανονικά ή παραδοσιακά αναπτύσσονταν από στρατιωτικές μονάδες. Μιλώ για παράδειγμα για το Μαλή. εκεί όπου έχουμε μια αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ποιος θα φυλάσει για παράδειγμα το στρατόπεδο. Μπορεί να το, κάνει, να το κάνουν και οι ίδιοι οι στρατιώτες, οι στρατιωτικές μονάδες. Αλλά θα μπορούσε πράγματι κανείς να πει ότι ναι, εδώ έχει νόημα να προσληφθεί ε, μια ιδιωτική εταιρεία ασφάλειας. Και γι' αυτόν τον σκοπό πράγματι ε, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο ώστε να μπορούν να γίνουν προσλήψεις από εδώ και όχι να πηγαίνουν οι εταιρείε εκεί και να προσλαμβάνουν κόσμο. Τώρα, για την για το επιχείρημα ότι ενδεχομένως πολλές φορές οι ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες ε, είναι σε θέση ή επιδιώκουν ενδεχομένως να κάνουν πράγματα τα οποία επίσημες κρατικές στρατιωτικές μονάδες δεν θα μπορούσαν. Αυτό για μένα είναι πραγματικά κόκκινη γραμμή. Εδώ θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες που θα ισχύουν για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι θα απαγορεύουν την διάπραξη, ε, την, ε, οι οποίες ε, δεν θα επιτρέπονταν ε, σε στρατιωτικές μονάδες να εκτελούνται από ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας. Ευχαριστώ. Κλείνω το κατάλογο των ομιλητών. Ο κύριος Φρόιντ είναι επόμενος. Ο κύριος Φρόιντ, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Φάτμεν. Πολλά υπόθηκαν ήδη από τους συναδέρφους και συμφωνώ, κυρίως με τον κύριο Μπούχνερ και την κυρία Τρικίενε. Και έχω να προσθέσω το Νομίζω ότι έχουμε εδώ ένα πρόβλημα που κινδυνεύει να βγάλει την υπόθεση αυτή, να τη χάσουμε από τα χέρια μας. Είναι αλήθεια ότι χρησιμοποιούμε αυτές τις ιδιωτικέ εταιρείε ασφάλειας χωρίς να τις ελέγχουμε. Αναφέρθηκε στην Blackwater, για παράδειγμα, ο κύριος Μπάχνερ, όπου έγιναν ε, από αυτήν παραβιάσεις φοβερές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην αρχή υπήρξε απόλυση, αλλά μετά όλα αυτά ξεχάστηκαν. Δεν θέλω βέβαια να αμφισβητήσω ότι είναι σημαντικό το έργο των εταιριών αυτό και δεν θέλω να τα βάλω όλα στο ίδιο καλά. Αλλά κυρία Βάτμεν, το γνωρίζετε, έχετε στοιχεία ε, καταχρήσεων που έχουν γίνει, που έχουν ξεφύγει από τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους άτομα που δουλεύουν για τις εταιρείες αυτές. Το προσωπικό πάντως, να ξέρετε, των εταιριών αυτών είναι από το πιο χαμηλοπληρωμένο που σημαίνει ότι οι ιδιωτικέ αυτές εταιρείες ασφάλειας είναι μεγάλη business και μάλλον γι' αυτό πολλαπλασιάζονται διεθνώς με τέτοιο ρυθμό. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο κύριος Κούκαν τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που συζητάμε το ζήτημα αυτό. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να ασχοληθούμε με το ζήτημα αυτό στη δική μας την υποεπιτροπή και προσβλέπω στο να καταλήξουμε σε μια κοινή τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το ζήτημα αυτό θέτει και ένα δίλημα, δηλαδή σε ποιο βαθμό ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας επιτρέπεται να αντικαταστήσουν το ρόλο των ίδιων των κρατών στην παροχή ασφάλειας. Το ζήτημα θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο και εκτιμώ ιδιαίτερα το πρώτο σχέδιο έκθεσης της εισηγήτριας που ασχολείται με τα πιο ουσιώδη ζητήματα που τίθενται με τις ιδιωτικέ εταιρείε ασφάλειας απαιτεί πιο συγκεκριμένε κατζήρε γραμμέ όσον αφορά την σύναψη συμβάσεων. Λέει θα πρέπει να υποβάλλονται εκθέσει και να καλυπτούν νομικά κενά, όπω λέγεται στην παράγραφο 16 συγκεκριμένα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όντω αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα συνεκτικό νομικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις εκτός χώρας προέλευσης. Πρέπει να δούμε όμως τι μορφή θα πρέπει να πάρει αυτό το κοινό νομικό πλαίσιο. Επίση, ασχολούμεθα με την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθότι οι ιδιωτικέ εταιρείε ασφάλειας χρησιμοποιούνται και σε στρατιωτικέ και μη στρατιωτικέ πολιτικέ προστασία, όπω άλλωστε ακούστηκε και στα πλαίσια της συζήτησης Και νομίζω ότι ε, όντω μπορούν να επηρεάσουν και τη δημόσια εικόνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω λέγεται στην παράγραφο 6 του σχεδίου έκθεση. Συνεπώ, είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα τη υφιστάμενη κατάσταση με τη δραστηριότητα των ε, ιδιωτικών αυτών εταιριών ασφάλεια. Και μια παρατήρηση τεχνική φύση ενδεχομένω θα ήταν θετικό να έχουμε περισσότερα δεδομένα που θα μπορούσαν να εμπλουτίσουν την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Και εμεί ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Νάατ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε για το ότι η θεμητή και δημοκρατική χρήση της ε, ισχύω είναι μονοπόλιο των χωρών μελών, της αστυνομίας ή των ενοπλών δυνάμεων. Ο δρόμος λοιπόν που έχουμε πάρει με φοβερή ταχύτητα μας ε, οδηγεί σε ε, ηθική καταβάθρωση οι χώρες δεν θέλουν να έχουν ε, νεκρούς στα πεδία της μάχης και χρησιμοποιούν είτε drones είτε μισθοφόρους. Ειλικρινά, θυμάμαι τον Μαρκ Χόλτ και άλλους, οι οποίοι τελικά τι κάνουν, παρέχουν υπηρεσίες σε περίπτωση ανάγκης, όχι, πρόκειται για μισθοφόρους. Πρέπει να διακρίνουμε λοιπόν τι σημαίνει η υλικοτεχνική ε, αρρωγή, κανείς δεν είναι κατά, και τι σημαίνει η πραγματικότητα ορισμένων ε, τέτοιων εταιριών, η Blackwater που μετά ονομάστηκε Academy και μετά δεν ξέρω εγώ πώς, ε, η Valcoms και άλλες, που αυτό που είναι, είναι απλώς μισθοφόροι που χρησιμοποιούν βαρύ οπλισμό στη Σιεραλεώνα, για παράδειγμα, σοβιετικά τάγκς και αυτό που κάνουμε είναι ότι εξάγουμε ένα πολιτικό ζήτημα, επειδή οι χώρε δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν δικούς τους στρατιώτες για τα αυτό εσωτερικά τους δημιουργεί πολιτικό ζήτημα, χρησιμοποιούν αυτού του μισθοφόρους. Αν πεθάνει ένα τέτοιο ε, υπάλληλο ιδιωτική εταιρεία δεν τρέχει τίποτα. Κι όμω στο άρθρο 1 του ψηφίσματο του ΟΗΕ, το λέει, μιλάμε για μισθοφόρους τους οποίους ονομάζουμε ιδιωτική εταιρεία ασφάλειας, ενώ αυτό που κάνουν είναι καθαρά στρατιωτικές επιχειρήσεις. Προσοχή λοιπόν. Η συμπεριφορά πρέπει να ανταποκρίνεται στη τόσα λέει Διεθνής Αμνηστία. Η Διεθνής Αμνηστία μίλησε για φοβερούς βασανισμούς στο Ιράκ και αλλού. Συνεπώς στηρίζω το ψήφισμα και πάνω απ' όλα τις τροπολογίες της Χίλντε, αλλά και τις δικές μου βέβαια, όπου μιλάω για την απαγόρευση παρουσίας των ιδιωτικών αυτών εταιριών ασφάλειας σε στρατιωτικές επιχειρήσεις σε εμπόλεμες περιοχές. Μιλάμε για μισθοφόρους και όχι για επιχειρήσεις ασφάλειας, που είναι μερικές φορές και εγκληματίες. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, όπως είπα και την αρχή, έχω και εγώ μια ερώτηση για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Γνωρίζουμε ότι ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας χρησιμοποιούνται στην Ουκρανία. Χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της ρωσικής επίθεσης κατά των ανατολικών εδαφών της Ουκρανίας. Στη Ρωσία υπάρχουν τουλάχιστον 10 ε, στρατιωτικές ε, δυνάμεις που δεν είναι αυθεντικές. Οι στρατιώτες τους χρησιμοποιήθηκαν στην Ουκρανία. Ρωτάω λοιπόν, δεν θα ήταν χρήσιμο να μιλήσουμε και γι' αυτό στην έκθεσή σας, να γίνει γνωστό, γιατί δεν το γνωρίζουν πολύ. Και τώρα, Χίλντε, έχεις το λόγο για να απαντήσεις στις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ όλους σας, συνάδελφοι, για τα όσα είπατε, όσα ζητήσατε. Σήμερα το πρωί ερχόμουν στις Βρυξέλλες, ευχόμουν να είναι όλοι οι ευρωβουλευτές εδώ στις 9 γιατί για μένα είναι μια πολύ σημαντική έκθεση και ήσασταν εδώ οπότε σας ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι πολύ για τις παρατηρήσεις σας και για τη στήριξή σας γιατί νομίζω ότι αυτή είναι η αίσθηση που δημιουργείται ότι υπάρχει ευρεία στήριξη και ότι όλοι λίγο πολύ ζητάτε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα και να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση που αναφέρω στην έκθεσή μου. Φυσικά πρέπει να υποβάλουμε και τροπολογίες να βελτιώσουμε το κείμενο, αλλά πάντα λέμε στο Βέλγιο μια συνάδελφος πολιτικός λέει τι, ότι όταν κάποιος είναι πάνω στο άλογο, το έχει καβαλήσει. Γίνεται κανείς πιο έξυπνος, επειδή είναι δύο κεφάλια που δουλεύουν, παρά όταν κάποιος δεν είναι πάνω στο άλογο. Έτσι λοιπόν και εγώ πιστεύω ότι με τη δικιά σας τη συνεργασία θα τα καταφέρουμε καλύτερα. Τώρα πολύ σύντομα κάποιες παρατηρήσεις. Για τόσο είπατε. Στην κυρία είπατε ότι χρειάζονται περισσότεροι κανόνες. Ναι, πράγματι, αυτό χρειάζεται. Περισσότεροι κανόνες για τους ένοπλους φύλακε και στη θάλασσα. Ναι, το λαμβάνουμε υπόψη. Το μονοπόλιο όμως του κράτους να χρησιμοποιεί βία υπάρχει. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η χρήση βίας είναι αρμοδιότητα των χωρών μελών. Αυτό είναι αλήθεια. Στον κύριο Φρουντζουλίκα. Πράγματι, πού είναι. Έφυγε. Ωραία. Λοιπόν, πρέπει να ρυθμίσουμε, πιστεύω, και το θέμα της συλλογή πληροφοριών από τις εταιρείε αυτές. Πράγματι, δύο-τρεις το είπατε. Δεν πρόκειται μόνο για οικονομικό ζήτημα. Όχι, δεν πρόκειται μόνο για οικονομικό ζήτημα. Για μένα το πιο σημαντικό, πιο σημαντικός λόγος για την έκθεση αυτή είναι να έχουμε περισσότερη ασφάλεια. Γιατί βλέπουμε ότι από μόνε του οι χώρε μέλη δεν τα καταφέρνουν. Και βλέπουμε ότι οι ιδιωτικέ αυτέ εταιρείε ασφάλεια δραστηριοποιούνται στον τομέα. Γι' αυτό και πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με την έκθεση αυτή. Στον κύριο Μπούχνερ τώρα. Μα στηρίζετε χοντρικά, είπατε ναι στην πράσινη βίβλο, οδηγία, ναι. Όλα όσα αναφέρατε, ναι, μιλάτε για τη δημοκρατική λογοδοσία, βεβαίως και υπάρχουν αυτά, εννοείται. Γι' αυτό και η έκθεση ζητάει ρυθμιστικό πλαίσιο, γιατί ακριβώς υπάρχουν παραβιάσεις. Το πιο σημαντικό για μένα είναι η ασφάλειά μας. Το οικονομικό μπορεί να είναι σημαντικό, αλλά η ασφάλεια δικιά μου των παιδιών μου είναι σημαντική. Και γι' αυτό συνέταξα την έκθεση αυτή. Και γι' αυτό την προωθώ. Και μόνο. Ζητάτε οδηγία. Ναι. Βεβαίω θα συμφωνήσω. Βεβαίω θα χρειαστούμε κάποια στιγμή οδηγία. Οπότε, ναι, συμφωνώ μαζί σα. Για τον κύριο Σαφάουζερ. Α, ναι, εκεί είσαστε. Λέτε ποια είναι η προσθεθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, λοιπόν, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολούμαστε με μια πολιτική άμυνας και ασφάλειας, έτσι. Αυτό πρέπει να προσθεθεί στη συζήτηση. Ήσασταν ο πιο αρνητικός από όσου πήραν το λόγο κατά της άμυνας, κατά της έκθεσης αυτής. Δεν συμφωνώ με τα σχόλιά σας. Είπατε ότι η έκθεση αυτή θα ιδιωτικοποιήσει τις ένοπλες δυνάμεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, δεν είναι αυτό ο στόχος της έκθεσης. Στόχος της έκθεσης είναι ότι χρειαζόμαστε περισσότερη ασφάλεια και οι ιδιωτικές εταιρείες ασφάλεια δραστηριοποιούνται, οπότε γι' αυτό και πρέπει να ασχοληθούμε. Οι επίσημες δυνάμεις, αν μας αν συνεργαστούν πιο στενά επιτόπου με ιδιωτικέ εταιρείε ασφάλεια και υπάρξει καλύτερη συνεργασία, τότε θα έχουμε καλύτερη και περισσότερη ασφάλεια. Αυτή είναι η άποψή μου. Και νομίζω ότι είναι Θετική επ' αυτού οι περισσότεροι συνάδελφοι. Αν θέλετε να τα πούμε οι δυο μας κάποια στιγμή, ελπίζω να σας πείσω. Κύριε Γκάλερ, τι αναθέτουμε στις ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας. Ε, την προστασία μας. Πράγματι αυτό είναι ένα από τα καθήκοντά τους. Και είπατε, δεν θα ήταν καλύτερα να έχουμε ένα θετικό κατάλογο αντί να έχουμε ένα μαύρο κατάλογο, μια μαύρη λίστα δεν είμαι πεπισμένη. Ίσως να πιούμε ένα καφέ μαζί και να προσπαθήσετε να με πείσετε. Γιατί αν κάνετε μόνο ένα θετικό κατάλογο, τότε κάνουμε μεγάλη χάρη στις μεγάλες εταιρείε και δεν θα βοηθήσουμε τις μικρότερες. Αυτή είναι η γνώμη μου. Αλλά ίσως μπορέσετε να με πείσετε για το αντίθετο. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη, γιατί ξέρω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο. Κύριε Φρόιντ, Ναι, ρωτάτε, έχουμε στοιχεία. Ναι, υπάρχουν ε, στοιχεία σε εθνικό επίπεδο και γι' αυτό και εμείς ζητούμε να τα έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κύριε Κούκαν, ε, θέσατε το σωστό ερώτημα. Περισσότερα στοιχεία. Ναι, αυτό το ζητάμε στην έκθεση. Κύριε Νάρ, αγαπητέ συνάδελφοι, χθε το συζητήσαμε και ευχαριστώ πολύ για τις καλές προτάσεις και τροπολογίες. Ξέρω ότι θα μας βοηθήσετε, θα βοηθήσετε την υποπιτροπή μας για μια καλή ισορροπία. Πρόεδρε, εσείς μου θέσατε το πιο δύσκολο ερώτημα. Κατά πόσο πρέπει να μιλήσουμε στην έκθεση αυτή για την Ουκρανία. Η πρώτη μου αντίδραση είναι όχι, γιατί δεν νομίζω ότι αυτό είναι ο κατάλληλο χώρο. Όμω, ναι, συμφωνώ ότι κάπου πρέπει να μιλήσουμε για την Ουκρανία. Οπότε ίσως μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στη συζήτηση, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να είναι ένα σημείο στην έκθεση. Αν όμως επιμένετε, θα πιω και μαζί σας ένα καφέ και θα προσπαθήσω... Ναι, όλοι μαζί θα πιούμε καφέ τελικά, εντάξει. Δεν ξέρω τι πιστεύουν οι υπόλοιποι. Νομίζω ότι είναι σημαντικό το θέμα αυτό που βάζετε το ότι πρέπει να το συζητάμε εδώ στην Επιτροπή μας, δεν ξέρω σε ποιο σημείο. Θα το αφήνω σε εσά, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν για τα θετικά σας σχόλια, συνάδελφοι. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πω ότι ο πόλεμος αυτός βρίσκεται στη γειτονιά μας. Πεθαίνουν άνθρωποι και πράγματι αξίζει να αναφερθεί κάπου. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτή την εξαιρετική συζήτηση. Κυρία Βάουτμαντ, σας ευχαριστούμε πολύ για την σύνταξη αυτού του σχεδίου έκθεσης που είναι πάρα πολύ χρήσιμη και πάρα πολύ σημαντική. Και με αυτό θα ήθελα να κλείσω το θέμα αυτό της ημερήσιας ε, διάταξης. Να σας υπενθυμίσω ότι η, υποβολή, η προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι η 16η Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και για την προσοχή σας, κυρία Φάουτμαντς. Και με αυτό περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, στο σημείο 5 there, there, Mrs. We, we give the floor first to Mrs. Gunslinger and then to Mrs. We bring them, we bring them up to the podium. Když dovolíte, otevřu bod číslo. Bod číslo. Λοιπόν, σημείο υπαριθμών 5 της ημερήσιας διάταξης. Στρατηγική εταιρική σχέση ε, ε, ΟΗΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιχειρήσεις διατήρηση Ειρήνης και Διαχείρισης Κρίσεων. Έχουμε δύο εξαίρετου προσκεκλημένους. Já bych Σας καλωσορίζω. Να πω ότι η εταιρική σχέση ΟΗΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργήθηκε το 2003 και βρισκόμαστε στο μέσο της εφαρμογής του σχεδίου δράσης ε, ε, που έχει καταρτιστεί ως προς την συμμετοχή ε, ευρωπαϊκών τμήματων και μονάδων ε, σε επιχειρήσεις του ΟΗΕ για τη διατήρηση της ειρήνης. Θα ήθελα λοιπόν να μας πούν οι ομιλήτριες που έχουμε σήμερα μαζί μας ε, ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή αυτού του σχεδίου δράσης. Πρώτο, πρώτη έχει το λόγο η κυρία Γκάνσλαντ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θέλω να τονίσω πόσο σημαντική είναι αυτή η στρατηγική εταιρική σχέση για τη διατήρηση της ειρήνης και την ε, διαχείριση των κρίσεων. Είναι μία από τις πιο θεμελιώδεις ε, εταιρικέ σχέσεις στον τομέα της, κοινων... της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο, σε πολύ καλό δρόμο ο οποίο χαράχτηκε τα προηγούμενα χρόνια και ακολουθούμε ε, τον δρόμο αυτόν. Στην ετήσια ε, συνάντηση ε, του Συμβουλίου Ασφαλείας τον Ιούνιο του 2016 αναδείχθηκε ο μοναδικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως εταίρος του ΟΗΕ σε διεθνή ζητήματα διατήρησης ειρήνης. Αυτή η συνεργασία Ενωμένων Εθνών και Ευρωπαϊκής Ένωση, στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας ωφελεί και τους δύο οργανισμούς και επικεντρωνόμαστε στα επιχειρησιακά ωφέλη επιτόπου. Η συνεργασία ε, με τον ΟΗΕ θέτει τις ε, αποστολές μας ε, εντός ενός ευρύτερου πολιτικού και στρατιωτικού πλαισίου που τις καθιστά πιο αποτελεσματικές αφενός, αλλά ταυτόχρονα συμβάλλει και στην ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση ε, της ε, πολυμερούς συνεργασίας. Τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω αυτής της στρατηγικής εταιρικής σχέσης ε, μοιράζονται τον φόρτο ε, των ε, αποστολών αυτών, όπως για παράδειγμα ε, οι αποστολές μας στην Κεντρική, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, στη Σομαλία, στο, στη Λιβύη, στο κέρας της Αφρικής και στην Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένα, η συνεργασία στους τομείς αυτούς εμπεριέχει τρία βασικά επίπεδα. Πρώτον, έχουμε έναν τακτικό διάλογο υψηλού επίπεδου συμπεριλαμβανομένης και της ε, Διοικούσας Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΗΕ που συνέρχεται δύο φορές τον χρόνο και τις οποίες προεδρεύει ο ε, αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σεράνο και ε, ο ομόλογος του από τον ΟΗΕ. Η επόμενη συνεδρίαση θα ε, πραγματοποιηθεί στις 16 Μαρτίου στη Νέα Υόρκη. Εκεί θα έχουμε την δυνατότητα να συζητήσουμε για την επιχειρησιακή συνεργασία και την επιτόπου συνεργασία, ιδίως στην Σομαλία, το Μαλί, τη Λιβύη και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και θα γίνει και ένας απολογισμός για την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σχέση με τη στρατηγική εταιρική σχέση ε, ΟΗΕ ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα έγγραφο που εγκρίθηκε ε, από τα κράτη-μέλη στην Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας. Και με αυτό περνάω στο δεύτερο επίπεδο, που είναι η κοινή στρατηγική εταιρική σχέση ΟΗΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης και διαχείρισης κρίσεων και οι προτεραιότητε που έχουν οριστεί για την περίοδο 15-18 και που εφαρμόζονται αυτή την περίοδο. Οι 7 τομεί προτεραιότητα που προσδιορίζονται σε αυτήν την ε, στρατηγική εταιρική σχέση περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την ταχεία ανταπόκριση, τη διευκόλυνση τη της ε, των κρατών μελών σε επιχειρήσεις διατήρησης τη ειρήνης του ΟΗΕ και τη συνεργασία ε, όσον αφορά την επιμελητία. Πέραν αυτών των τομέων, Σημαντικά θέματα που μας απασχολούν είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ανάπτυξη, ε, όπου επίσης γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων με τον ΟΗΕ. Η συνεργασία περιλαμβάνει και το συντονισμό επιτόπου, καθώς και ανταλλαγές απόψεων και πληροφοριών μεταξύ ε, στρατηγικών ε, μονάδων όσον αφορά τι εντολές. Και αυτές οι ανταλλαγέ είναι πάρα πολύ σημαντικές όσον αφορά την αποτελεσματική συνεργασία επιτόπου, καθώς ε, βοηθούν στον εξορθολογισμό της διεκπαιρέωσης των καθηκόντων και βοηθούν, συμβάλλουν στην επίλυση προβλημάτων και διευκολύνουν την συνεργασία Η συνεργασία μεταξύ των αποστολών μας επιτόπου επίσης περιλαμβάνει την αμοιβαία υποστήριξη, όπου ε, ε αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ εξυπηρετούν οι μεν της δε ε, στον τομέα της ε, φιλοξενίας, της στέγασης, ε, της παροχής ιατρικών υπηρεσιών. Είναι πολύ σημαντική η συνεργασία αυτή για την συνεργασία και την εφαρμογή των εντολών των αποστολών μας. Έχω κάποια παραδείγματα συνεργασία τα οποία θα μπορούσα να σα δώσω, αλλά νομίζω ότι καλό θα ήταν να σταματήσω εδώ και να επανέλθω σε αυτά τα παραδείγματα, αν και εφόσον υπάρχουν και σχετικέ ερωτήσει. Αν συμφωνείτε κι εσεί, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Όντω, καλύτερα να προχωρήσουμε έτσι. Να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Άννη Χέντς η οποία είναι αναπληρώτρια προϊστάμενη του Γραφείου Σύνδεσης των Ηνωμένων Εθνών για την Ειρήνη και την Ασφάλεια. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας να μιλήσω εδώ στην Επιτροπή σας Άμυνας και Ασφάλειας όσον αφορά την στρατηγική ιδερική σχέση Ηνωμένων Εθνών και Ευρωπαϊκή Ένωση, επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης και διαχείριση κρίσεων. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλώ μετά την κυρία Κλάρα Γκάνσλαντ, με την οποία συνεργάζομαι σε τακτικό καθημερινό επίπεδο. Όντω εργάζομαι στο Γραφείο Σύνδεση των Εθνών για την Ειρήνη και την Ασφάλεια. Πρόκειται για, μια, ένα γραφείο το οποίο ασχολείται τόσο με πολιτικές υποθέσεις όσο και με ειρηνευτικές επιχειρήσει δημιουργήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Εθνών το 2011 προκειμένου να προωθηθεί εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε στήματα ειρήνη και ασφάλεια. Το UNLOPS λοιπόν επικεντρώνεται στο συντονισμό, το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή επιχειρήσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των εθνών με συντονισμό πολιτική, γενική παρακολούθηση και υποβολή ε, εκθέσεων όσον αφορά τι επιχειρήσει διατήρηση τη Ειρηνή και διαχείριση κρίσεων. Η Κλάρα αναφέρθηκε πριν από λίγο σε έναν όργανο που έχει δημιουργηθεί, την Steering Committee, τη Διευθύνουσα Επιτροπή όσον αφορά τη διαχείριση των κρίσεων. Έχουμε επίση τον θεσμικό διάλογο και προβλέπονται οι μερίδε επίλυση διενέξεων στο τέλο του μήνα στι Βρυξέλλε. Και επίση έχουμε και την άτυπη ομάδα φίλων, η οποία συνεδριάζει στι Βρυξέλλε κατά περίπτωση. Θα γνωρίζετε το έργο των ΗΕ, Εθνών. Για να σας πω πολύ σύντομα όμως πώς λειτουργούν τα πράγματα. Το γραφείο αυτό ε, πολιτικών υποθέσεων καθώς επίσης και το γραφείο ε, επίλυσης ε, κρίσεων λειτουργεί στην Νέα Υόρκη. Έχουμε, διεξάγουμε 42 ειρηνευτικέ διαδικασίε, εκ των οποίων επιχειρήσει με συγχωρείτε, 17 εκ των οποίων είναι επιχειρήσει διατήρηση τη Ειρηνή, ενώ 25 είναι πολιτικέ αποστολέ και αποστολέ καλών υπηρεσιών. Απασχολούμε περίπου 130.000 προσωπικό παγκοσμίω, 90.000 στρατιώτε, 13.500 αστυνομικό προσωπικό και περίπου 2.000 στρατιωτικού παρατηρητέ ο συνολικό μα προπολογισμό υπερβαίνει τα 9 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίω. Όπω είπε και η Κλάρα, η εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντική. Ο γενικό μα Γραμματέα τον αγνωρίζει αυτό και μάλιστα στι 21 Φεβρουαρίου στην ανοιχτή συζήτηση που έγινε στο Συμβούλιο ασφαλεία για την επίλυση κρίσεων με τη συμμετοχή εκπροσώπων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Γενικό Γραμματέας εκτίμησε ιδιαίτερα την εργασία που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την πρόληψη διενέξεων και συγκρούσεων και όντως ε, συνεργαζόμαστε παράλληλα με αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κεντροφρεκανική Δημοκρατία, στο Μαλί, τη Σομαλία, τη Λιβύη και στη Μέση Ανατολή. Είμαστε λοιπόν παρόντες ε, σε κάποιες από τις πιο σημαντικές διενέξεις. Η Κλάρα κάλεψε το πλαίσιο πολιτικής καθώς επίσης και τις κοινέ μας δράσεις στα πλαίσια της στρατηγικής αυτής εταιρικής σχέσης ΗΕ και Ευρωπαϊκής Ένωσης και για το παρόν και για τη μελλοντική περίοδο και να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση που έχει κάνει τη δικασία πραγματικά κοινή και λειτουργεί υπέρ τόσο τη Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και των ΗΕ και ξέρω ότι η Κλάρα θα περάσει σε κάποιες πρακτικές λεπτομέρειες όσον αφορά την συνεργασία αυτή. Θα ήθελα εγώ με τη σειρά μου να αναφερθώ στον τρόπο συντονισμού Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Εθνών για τον σχεδιασμό των αποστολών μη στρατιωτικών και στρατιωτικών που είχαμε ήδη αρχίσει να εφαρμόζουμε στα πλαίσια της προηγούμενης στρατηγικής εταιρικής σχέσης στην κεντροφρακανική δημοκρατία, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποίησε την αποστολή γεφύρωσης το 2013 στην κεντροφροκανική λοιπόν δημοκρατία και έχουμε πλέον προτεραιότητες για την περίοδο 2015 με 2018 στα πλαίσια των οποίων θα έχουμε ένα κοινό σχεδιασμό ταχείας αντίδρασης και ανταπόκρισης και επίσης θα έχουμε και κάποιες συγκεκριμένε ασκήσεις προκειμένου να βιστοποιήσουμε περισσότερο το προσωπικό των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνών για το πώς θα μπορούν όντως να αντιδρούν γρήγορα στα πλαίσια τέτοιων ε, επιχειρήσεων ταχείας ανταπόκρισης. Όσον αφορά κάποιες άλλες μορφές πρακτικής συνεργασίας, να αναφερθώ σε κάποια πράγματα πολύ γρήγορα, τα βλέπετε και στις διαφάνειες. Αναφέρθηκα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Έγινε μία αναθεώρηση μετά την συνεργασία αυτή, μετά την επιχείρηση αυτή. Και επίσης να σας πω ότι είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Μαλί, ιδίω στα πλαίσια του κοινού πλαισίου αμοιβαίας υποστήριξης και ιδίω στα πλαίσια των ενεξελίξη προσπαθειών η Μινούσμα να υποδεχθεί την EUTM στο Γκάο, στα βόρεια της χώρας, Πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό προκειμένου να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε κάποιες από τις μεγάλες προκλήσεις που πλήττουν ε, τη χώρα αυτή σε μια κατάσταση η οποία όλο και επιδεινώνεται. Αξιότιμα λοιπόν μέλη, θα ήθελα επίσης ε, να σας ε, πω πώς έχουν τα πράγματα όσον αφορά τις εξελίξεις των ΟΕΕ στον τομέα της ειρήνης και της ασφάλειας. Ξέρετε ότι προσπαθούμε να τροποποιήσουμε την προσέγγιση μας κατά τρόπο σημαντικό. Έγινε μια αναθεώρηση λοιπόν το 2015, η Peace Operation Review, την γνωρίζετε ως HIPPO, H-I-P-P-O. Ήμουνα 6 μηνών, 7 μηνών έγκυος όταν χρειάστηκε να κάνω την παρουσίαση αυτή και τη HIPPO. Είναι το ανεξάρτητο βαθμό πάνελ για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις. Στα πλαίσια της σημαντικής λοιπόν αυτής αναθεώρησης Μιλήσαμε πάρα πολύ για τις εταιρικέ σχέσεις. Γι' αυτό το λόγο το δικό μας το γραφείο στα Έθνη έχει αναλάβει όλο και σημαντικότερο ρόλο στα πλαίσια της Γενικής Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών, ακριβώς επειδή συνειδητοποιούμε ότι θα πρέπει να έχουμε πιο στενή εταιρική σχέση με εταίρους όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση καθότι αυτό μπορεί να συμβάλλει πάρα πολύ στην εδραίωση της ειρήνης, στην πρόληψη των συγκρούσεων και επίσης μπορούμε να βελτιώσουμε κατά αυτόν τον τρόπο το σχεδιασμό αλλά και την ίδια την εξαγωγή των ειρηνευτικών αποστολών. Η εταιρική σχέση είναι δύσκολο πράγμα και τα Ηνωμένα Έθνη είναι μια τεράστια, όπως ξέρετε, γραφειοκρατία, το ίδιο βέβαια και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ένας τεράστιος γραφειοκρατικός θεσμός. Προσπαθούμε λοιπόν να κινητοποιηθούμε και να οργανωθούμε εσωτερικά προτού ανοιχτούμε προ τα έξω. Από πρακτική πλευρά λοιπόν τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά και από πολιτική πλευρά είναι δύσκολα. Γιατί στην πράξη μια άλλη οντότητα πέρα από τα Ηνωμένα Έθνη και αυτό μπορεί να σοκάρει λίγο τους συναδέλφους στη Νέα Υόρκη. Παραδεχόμαστε ουσιαστικά ότι κάποιοι μπορούν να είναι πιο αποτελεσματικοί από εμά. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει ότι είναι πάρα πολύ αποτελεσματική στην παροχή εξειδικευμένων ικανοτήτων, καθώς επίσης και στα πλαίσια της μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, μέσω της Άμισομ επίσης στο Μαλί η Αφρικανική Ένωση με τη σειρά της έχει δείξει ότι μπορεί να συμβάλλει πολύ περισσότερο στην καταπολέμηση των εξεγέρσεων και στην εδραίωση της ειρήνης περισσότερο από την ΟΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν και η Αφρικανική Ένωση είναι πολύ σημαντικοί εταίροι οι οποίοι πραγματικά μπορούν να προσφέρουν εμόχλευση μεγαλύτερη από αυτή που μπορεί να προσφέρουν τα ενωμένα Έθνη. Τα ενωμένα Έθνη μπορούν να συμβάλλουν με τη σειρά του χρηματοδοτικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση όμω μπορεί να γνωρίζει καλύτερα πώ έχουν τα πράγματα σε μια χώρα, ενώ η Αφρικανική Ένωση έχει πολλέ φορέ δυνάμει επιτόπου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι οι τρεις πυλώνες της αναθεώρησης των ειρηνευτικών επιχειρήσεων προβλέπουν ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα πρέπει να συμβάλλουν στην πολιτική διευθέτηση των διενέξεων και δεν θα πρέπει αυτές να παγώνουν επί τόπου. Ο καθένας από τους πυλώνες αυτούς της αναθεώρησης που του ονομάζουμε 3P στα αγγλικά, εταιρική σχέση, σχεδιασμός και πρόληψη, περιέχουν πάρα πολλές συστάσεις. Και η Γενική Γραμματεία παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις 94 αυτές συγκεκριμένες συστάσεις, δράσεις αν θέλετε, τις οποίες δεν θα σας παρουσιάσω τώρα την κάθε μία ξεχωριστά. Θα ήθελα απλώς να αναφερθώ σύντομα στο λόγο για τον οποίο τα Ηνωμένα προχώρησαν σε αυτόν τον δρόμο. Γιατί και οι επιπτώσεις είναι σημαντικές και για μας. Οι εμφύλοι πόλοι έχουν τριπλασιαστεί τελευταία χρόνια. 125 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια. 60 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους και ένα 80% των υφιστάμενων ανθρωπιστικών αναγκών προκύπτουν από βίες, διενέξεις και συγκρούσεις. Το οικονομικό κόστος λοιπόν των διενέξεων αυτών θα ξεπερνάει αυτή τη στιγμή τα 14-3 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Επίσης οι διενέξεις αυτές είναι πολύ πιο πολύπλοκες επηρεάζουν μία την άλλη, ξεπερνούν πολλέ φορέ τα εθνικά σύνορα, επεκτείνονται σε ολόκληρε περιφέρειες, οδηγούν σε ριζοσπαστικοποίηση, σε βίο εξτρεμισμό και θέτουν συγκεκριμένε προκλήσει για την παγκόσμια ασφάλεια. Αυτό το είδαμε για παράδειγμα στην επιδείνωση τη κατάσταση που έχουμε στη Συρία και στην Ιεμένη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ποιε είναι οι επιπτώσει τη δική μα αποτυχία να, να προλάβουμε τι κρίσει αυτέ Και τονίζω τον όρο αποτυχία η διεθνής κοινότητα και την Ηνωμένα Έθνη έχουν αποτύχει αυτή τη στιγμή σε χώρες όπως η Συρία. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του επιδεινόμενου διεθνούς πλαισίου κάναμε την αναθεώρηση της στρατηγικής μας. Ο στόχος της αναθεώρησης αυτής της Γενικής Γραμματείας ήταν να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε τα Ηνωμένα Έθνη πιο αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Επίσης υπάρχουν και κάποιες επιχειρησιακές εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας που είναι σημαντικές και που άρχισαν να λαμβάνουν χώρα το 2015 και που επηρέασαν την αναθεώρηση της στρατηγικής μας. Καταρχάς έχουμε πολλές νέες καινοτομίες όσον αφορά τις ρενευτικές επιχειρήσεις. Έχουμε τις τρεις κλασικές φάσεις επιχειρήσεις αυτές, η παρακολούθηση για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή έχουμε αυξήσει τα καθήκοντα αυτά. Έχουμε φτάσει τα 40 καθήκοντα, έχουμε και προστασία ακόμα και τον, του άμαχου πληθυσμού. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όντω η στρατηγική μας αυτή περιπλέκεται. Είχαμε όμως και άλλες επιχειρήσεις ειρηνευτικές για την καταπολέμηση του εμπόλα, για παράδειγμα, ή η κοινή επιχείρηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την, τον περιορισμό των χημικών όπλων. Βλέπουμε επίση ότι ε, υπάρχουν, υπάρχει όλο και μεγαλύτερη συμβολή από την Αφρικανική Ένωση, για παράδειγμα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και στο Μαλί. Επίση βλέπουμε ότι υπάρχουν όλο και περισσότερε πρωτοβουλίε εδραίωση και διατήρηση τη ε, ειρήνη παγκοσμίω. Και αυτό περιπλέκει κάπω τα πράγματα. Στα δύο Σουδάν, και αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον, έχουμε δέκα εντεταλμένου και διαμεσολαβητέ από πέντε διαφορετικά θεσμικά όργανα πέρα από τις τρεις επίσημες αποστολές των Ηνωμένων Εθνών. Και επίσης βλέπουμε ότι το προσωπικό μας στις αποστολές αυτές κινδυνεύει όλο και περισσότερο καθότι συμμετέχει σε διενέξεις υψηλής έντασης στην κεντροαφρικανική δημοκρατία, στην Αλλαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, στο Μαλί, αλλά τελευταία και στα υψίπεδα Γκολάν. Να αναφερθώ τώρα εν συντομία και στον τρόπο εφαρμογή τη στρατηγική μα και τη εταιρική σχέση, γιατί αυτό είναι εξίσου σημαντικό. Έχουμε 94 συγκεκριμένε δράσει, πολλέ εκ των οποίων βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην άμεση διοίκηση τη γραμματείας, άλλε βρίσκονται υπό τη διοίκηση των μελών των κρατών μελών του ΗΕ, ο νέο Γενικό Γραμματέα ο Αντώνιο Γκουτέρε είναι ένα ευρωπαϊο πολιτικό βέβαια και αυτό βοηθά πάρα πολύ τη συνεργασία μεταξύ ΗΕ και Ευρωπαϊκή Ένωση και ζήτησε να γίνει μια εσωτερική αναθεώρηση όσον αφορά την πιθανή αναδιάρθρωση της Γενική Γραμματεία για την άμυνα και την ασφάλεια. αποτελείται να τα γνωρίζουμε τον Ιούνιο του 2017 καθώς συζητάμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον πολιτικό διάλογο αντιμετώπιση τρομοκρατία, ο Γενικός Γραμματέας πρότεινε να δημιουργηθεί ένα νέο γραφείο για την καταπολέμηση τρομοκρατίας. Επίσης, ως Ηνωμένα Έθνη, καταφέραμε στον τομέα της πρόληψης να κάνουμε κάποια σημαντικά πράγματα. Έχουμε δημιουργήσει περιφερειακές, περιφερειακά γραφεία. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η περιφερειακή αυτή παρουσία, για παράδειγμα στη Δυτική Αφρική, την Κεντρική Ασία και την Κεντρική Αφρική, όσον αφορά τις ικανότητες σχεδιασμού. Έχουμε δημιουργήσει ήδη ένα γραφείο και ακολουθούμε ως μοντέλο την CNDB στα πλαίσια του εκτελεστικού γραφείου της Γενικής Γραμματείας το ζήτημα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης ε, αποτελεί βασική μας προτεραιότητα και το αντιμετωπίζουμε και αυτό στα πλαίσια της αναθεώρησης. Έχουμε μία προσέγγιση, μία πολιτική μηδενική ανοχής. Έχουμε συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης στα πλαίσια των ε, ε, στρατιωτικών αυτών επιχειρήσεων και αποστολών. Τώρα, πώς κινούμεθα στο μέλλον. Πρόληψη καταρχάς και διαμεσολάβηση. Οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να αποταλήσουν τμήμα του βασικού προπολογισμού των ΗΕ και χαιρόμαστε πάρα πολύ που η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του μέσου σταθερότητας και ανάπτυξης συμβάλλει στι προσπάθειε διαμεσολάβηση των ΗΕ. Αυτό θα πρέπει να αποτελέσει όμω μόνιμο στοιχείο του προπολογισμού των ΗΕ και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λάβουν υπόψη του την πρότασή μα αυτήν. Όπω σα είπα, συνεργαζόμαστε εκ του σύνεγγυ με την Ευρωπαϊκή Ένωση και στα πλαίσια των Conflict Prevention Days που θα λάβουν χώρα στο τέλος του μήνα στις Βρυξέλλες. Έχουμε επίσης και μια πρωτοβουλία όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, την οποία προωθούμε στα πλαίσια της Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να έχουμε κάποιες ε, ομάδες των ε, Ηνωμένων Εθνών στα πλαίσια των αποστολών εκείνων όπου είμαστε παρόντες για να έχουμε καλύτερη διευθέτηση των ε, διενέξεων, η αποφυγή, η πρόληψη των μελλοντικών διενέξεων. Επίσης θέλουμε να συνεργαζόμαστε περισσότερο με το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να έχουμε καλύτερη παρακολούθηση της δραστηριότητας της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας και επίσης θέλουμε να μπορούμε να χρηματοδοτούμε και να στηρίζουμε καλύτερα τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις της Αφρικανικής Ένωσης και καθότι συμβάλλει βέβαια σε επιχειρήσει αυτέ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πολύ σημαντικό να συνομιλούμε μαζί τη για να δούμε πώ μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε τι αποστολέ αυτέ. Συμμετέχουμε επίση περισσότερο στην Steering Committee της, για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Τώρα, τι επιφυλάσσει το μέλλον Όσον αφορά την ταχύη ανταπόκριση, αυτό θα συνεχίσει να αποτελεί μια πολύ σημαντική πτυχή της στρατηγικής μα σχέση. Είδαμε ότι λειτουργεί πολύ καλά το σύστημα, ότι συμβάλλει, συμβάλλει πολύ καλά η Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι συμβάλλει όντω στην εδραίωση τη σταθερότητα και τη ανάπτυξη και ότι μπορεί επίση να κινήσει περισσότερε μάχημε μονάδε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν να συμβάλλουν για την χρηματοοικονομική παρακολούθηση των αποστολών και εσείς μπορείτε από πολιτικής πλευράς να συμβάλλετε αποτελεσματικά και αναφέρομαι στο ψήφισμα αυτό το οποίο εγκρίνεται τον Ιούνιο του 2016 όσον αφορά την υποστήριξη των ειρηνευτικών αποστολών. Εκτιμούμε πάρα πολύ λοιπόν τη συμβολή σας αυτήν και καθώς επικεντρωνόμαστε όλο και περισσότερο στην πρόληψη στα Ηνωμένα Έθνη, μπορούν όντως ε, οι ευρωβουλευτές να συμβάλλουν πάρα πολύ στα πλαίσια της διαμεσολάβησης, ιδίως όσον αφορά τις αποστολές παρακολούθησης των εκλογών. Μπορούμε και εκεί λοιπόν να συνεργαστούμε περισσότερο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και τις δύο ομιλήτριές μας. Έχω να κάνω την εξής πρόταση. Σας κάνουμε δύο γύρους ερωταπαντήσεων. Πρώτος γύρος είναι ο κύριος Γκάλαρ, Λέζινγκ, Άναρ. Μετά τον πρώτο γύρο θα περάσουμε στο δεύτερο γύρο. Κύριε Γκάλαρ, λοιπόν, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις παρουσιάσεις αυτές. Είναι σημαντικό να σχηματίσουμε μια εικόνα για το πού υπάρχουν δυνατότητες και σε ποιους τομείς είναι σωστό και ενδεδειγμένο να υπάρχει μια θεσμική συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΟΗΕ. Και αν υπάρχουν καθιερωμένες δομές του ΟΗΕ, φυσικά είναι λογικό και σωστό να συνεισφέρουμε και εμείς σε αυτές. Εγώ δεν αμφισβητώ καμία από τις δραστηριότητες που αναπτύσσουμε από κοινού. Είναι σαφές αυτό. Αυτό που με απασχολεί είναι να γίνουν ορατές οι δραστηριότητες της, Ευ... της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ένα από τα πλέον ε, μακροχρόνια προβλήματα. Δίνουμε χρήματα, παρέχουμε προσωπικό και παρόλα αυτά ε, οι υπόλοιποι εν τέλει καταλήγουν να μας αντιλαμβάνονται ως αποστολή του ΟΗΕ και όχι ως αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι σημαντικό και θα ήθελα να καλέσω την Ευρωπαϊκή ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να εξασφαλίζει ότι η σημαία και τα εμβλήματά μας είναι πάντοτε ορατά. Δεν λέω ε, εκεί όπου ενδεχομένως υπάρχουν λόγοι που ε, δεν θα πρέπει να είμαστε στο προσκήνιο να το κάνουμε οπωσδήποτε. Παρόλα αυτά όμως νομίζω ότι είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η προβολή της παρουσίας και της συμμετοχής μας σε αυτές τις αποστολές και θα ήθελα να μου δώσετε ορισμένες πληροφορίες αν έχετε για το ποια είναι ακριβώς η κατάσταση επιτόπου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκάλερ. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπατε. Πιστεύω και εγώ ότι χρειάζεται να γίνουμε πιο ορατοί, να προβάλλεται περισσότερο η παρουσία μας και η συμμετοχή μας. Η κυρία Λέζινγκ, ευχαριστώ πολύ. Στις πρώτες ε, διαφάνειες ε, συμπεριλάβατε το αίτημα για τη διεύρυνση αυτής της ε, εταιρικής σχέσης ΟΗΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά τις ε, αποστολές της κοινή πολιτικής ε, ασφάλειας και άμυνας, από ό,τι καταλαβαίνω, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι περισσότερο συμπληρωματικός, υποστηρικτικός στις ε, αποστολές του, των Ηνωμένων Εθνών. Το ερώτημά μου είναι, καθώς μιλούμε κυρίως για χώρες του, του Νότου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει σε αυτές τις αποστολές. Υποστηρίζει με πόρους τις αποστολής, τις αποστολές αυτές επαρκώς για το, για το ζήτημα των African Peace Facilities. Υπάρχει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία έχει ασκηθεί έντονη κριτική στην κοινή γνώμη δημοσιογράφοι μου έχουν θέσει πολλάκις το ερώτημα πώς είναι δυνατόν ε, να χρηματοδοτούνται στρατιωτικές αποστολές με χρήματα και κονδύλια τα οποία ε, προβλέπονται και προορίζονται για ανθρωπιστική βοήθεια ή για αναπτυξιακή βοήθεια. Είναι και αυτό ένα θέμα που είναι απαραίτητο να συζητηθεί και εδώ στην Επιτροπή μας αλλά και στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Βαλέρο έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις σας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Έχω κάποιες ερωτήσεις Κοιτάξαμε κάποια έγγραφα εν ώψη της συνεδρίασης αυτής και εγώ θέλω να ξέρω περισσότερα για τον αριθμό των Ευρωπαίων πολιτών, πόσοι δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχουν σε παρεμβάσεις του Ηνωμένου Εθνών. 40.000 κάτι είναι το νούμερο που έχω βρει εδώ. 9.000 δεν είναι ένα μικρό νούμερο έτσι καλλιώς. Και εγώ είμαι από την Σουηδία. Σκέφτομαι ποιο είναι το πλαίσιο εκεί. Και ξέρω ότι στην ΙΣΑΦ έχουμε 600 που συμμετέχουν. Και όσον αφορά τις παρεμβάσεις του ΟΗΕ, αυτού καθ' αυτού, έχουμε 20 οι οποίοι πήγαν επί τόπου. Και πρόκειται για απευθείας δηλαδή δράσεις του ΟΗΕ. Οπότε θέλω να ξέρω, πρόκειται για άτομα τα οποία υπάγονται στον ΟΗΕ ή συμπεριλαμβάνονται και άτομα τα οποία δουλεύουν σε άλλες αποστολές υπό μια γενική εντολή του ΟΗΕ. Ποια είναι δηλαδή η πραγματικότητα πίσω από τα νούμερα αυτά. Έπειτα έχω μια άλλη ερώτηση. Για αυτά που ακούμε για τις μάχημες μονάδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι θα συμπεριλαμβάνονται δεχομένως και αυτές στις ε, επιχειρήσεις του ΟΙΕ. Και να ρωτήσω και κάτι και για μια επιχείρηση η οποία ήδη λαμβάνει χώρα με νοσού στη Δυτική Σαχάρα. Δεν συμβαίνει τίποτα εκεί. Οπότε τι γίνεται. Γιατί υπάρχει. Δεν υπάρχει καμιά πρόοδος. Οπότε Πώς θα αντιδρούσατε. Είναι μια επιχείρηση, θέλω να πω, που δεν έχει καταλήξει πουθενά. Δεν έχει φέρει αποτελέσματα. Δυστυχώ συμβαίνει αυτό. Που και που. Έχει να κάνει και με την αντίδραση των ευρωπαϊκών χωρών. Γιατί θέλουν να προστατεύσουν τις ανθρώπινες ζωές σε αυτό το σημείο του κόσμου. Αυτά προς το παρόν. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, Ευχαριστούμε. Ο κύριος ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ. Πραγματικά βρίσκω σκανδαλώδη κάποια από αυτά που άκουσα. Ο πόλεμος είναι πάρα πολύ σημαντικός για το να αφήνουμε στους στρατιωτικούς. Υπάρχει μια τέτοια ρίση. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό ισχύει για τους πολιτικούς. Όταν μιλάτε για τις σοβαρές επιπτώσεις της συνεργασίας ε, του ΟΙΕ με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε διάφορα σημεία του κόσμου, δεν ξέρω για ποια σημεία του κόσμου αναφέρεστε γιατί εκεί που πήγα εγώ, πήγα όχι μόνο κοιτώντα χαρτιά, αλλά βλέποντα την κατάσταση επιτόπου. Εδώ και τέσσερα χρόνια λοιπόν υπήρξε η αποστολή να ετοιμαστούν έξι τάγματα στο Μαλί. Θα το ξέρετε, και δεν ξέρω γιατί δεν μας το λέτε, ότι καμιά από τις μονάδες αυτές δεν λειτουργεί σε κανένα επίπεδο, ούτε καν 30 άντρες. Όταν λοιπόν μιλάτε για τους ε, ανθρώπους από την Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίοι εκπαιδεύουν, τι εκπαιδεύουν. Δέκα άντρε σε θέματα ασφάλειας. Είναι όμως μονάδες αυτές οι οποίες δεν λειτουργούν και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τους δίνει ούτε εξοπλισμό, ούτε καν το κάνει αυτό στο στρατό του Μαλή. Και όταν υπάρχουν μάχες, ε, φεύγουν, γιατί δεν μπορούν να μηνθούν. Όταν λοιπόν υλοποιείται μία επιχείρηση για να εκπαιδευτεί έξι τάγματα και καταλήγουμε σε 30 άντρε, αυτό είναι μια τεράστια αποτυχία. Και δεν μπορεί να μιλάμε για εξαίρετη συνεργασία και τι ωραίε που είναι οι σχέσει των ΗΠΑ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πήγατε εκεί για να συμπληρώσετε χαρτιά, αλλά για να εκπαιδεύσετε έξι τάγματα και κανένα από αυτά δεν χρησιμοποιείται. Δεν λειτουργεί. Έπειτα, η αντιπαράθεση επιτόπου με τα Ηνωμένα Έθνη. Σίγουρα θα έχετε δει αυτή την ε, ταινία. Ξενοδοχείο Ρουάντα, έτσι λέγεται. Ε, λοιπόν, τα όσα περιγράφονται εκεί είναι καθημερινή πραγματικότητα. Στο Σουδάν βλέπουμε τις φαγές που γίνονται των μεν κατά τον δε. Όταν μιλάμε για την εξαιρετική αποστολή στην Κεντροαφρικανική Ένωση, στον Πακί, έξω από τον Πακί, υπάρχει δάσος και γίνονται σφαγές από παραστρατιωτικούς. Λοιπόν, δεν μπορεί να ερχόσαστε εδώ και να μας εξηγείτε ποιες είναι οι αποστολές επιχειρήσεις που υπάρχουν και τι ωραία που υπάρχει ε, ταχεία αντίδραση. Μα δεν είναι ταχεία αντίδραση, αυτό είναι οξύμορο. Πήγα στο Κιντάλ, έτσι, που είναι εμπόλεμη η περιοχή. Όταν πήγα λοιπόν εκεί, τα δύο στοιχεία των του Άρεκ, η πλατφόρμα και ο συντονισμός, συνεργαζόντουσαν αποτελεσματικά, ενώ ο ΙΕ στην περίμετρο του Κεντάλ είχε κατακαιρματισμένες τις δυνάμεις του. Τελικά υπάρχει απαγόρευση δράσης σε βάθος. Όταν λοιπόν συζητάει κανείς με τους στρατιωτικούς όμως, έτσι, όχι με τους πολιτικούς, με αυτούς που όντως κάνουν τις επιχειρήσεις επιτόπου, με τους στρατιώτες που υποφέρουν, που πεθαίνουν, με τους αξιωματικούς, σας λένε ότι πρόκειται για αποτυχία, ότι δεν λειτουργεί, ότι δεν είναι επιχειρησιακή, ότι δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν οι τρομοκράτε επιτόπου. Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε ότι μερικές φορές στην έρημο κάποιος πρέπει να πάει 150-200 χιλιόμετρα. Σας το λέω ειλικρινά. Η αίσθηση που έχουμε, και θα ολοκληρώσω με αυτό, είναι πλήρους αποτυχίας. Ότι σε χαρτιά μόνο αναφέρονται αυτά που δεν είναι πραγματικότητα. Πρέπει να πάτε να μιλήσετε με αυτούς που βρίσκονται επί τόπου, με τους αξιωματικούς, με τους στρατιωτικούς του ΟΗΕ και με αυτού να μιλήσετε και με αυτού τη Ευρωπαϊκή Ένωση που ντρέπονται γιατί τελικά δεν μπορούν να προσφέρουν την εκπαίδευση που θα έπρεπε να προσφέρουν. Αυτή η εξωτερική συνεργασία που λέτε εσεί έχει καταλήξει σε τέσσερα χρόνια να μην έχουν εκπαιδευτεί ούτε 30 άντρε. Είναι τρομερή αποτυχία αυτό. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Ναρτέ. Ήσασταν ο τελευταίος στον κατάλογο ομιλητών στον πρώτο γύρο, οπότε τώρα θα ζητήσω από τις προσκεκλημένες μας να απαντήσουν. Στη συνέχεια θα περάσουμε σε δεύτερο γύρο. Προς το παρόν είναι ο κύριος Σαπφόιζερ στο δεύτερο γύρο. Λοιπόν, παρακαλώ κύριε Κάτσλα, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Και ευχαριστώ πολύ για όλες αυτές τις τόσο σημαντικές ερωτήσεις και τα σχολιά σας. Αρχίζω με το τελευταίο. Είμαι πεπισμένη ότι όλοι μπορούμε να μιλήσουμε για αποτυχία, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή σήμερα δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει εξοπλισμό για στρατιωτικές δράσεις. Η υπηρεσία εξωτερικής δράσης, οι χώρες μέλη το ξέρουν, όλοι μας. Και είναι ένα περίπλοκο ζήτημα. και συζητιέται και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Να εξεταστεί αυτή η νομοθετική πρόταση, δηλαδή με τροποποίησης τα εργαλεία που διαθέτουμε για την ε, σταθερότητα και την ειρήνη. Κάποιες λοιπόν από αυτές τις ανάγκες θα μπορούσαν να καλυφθούν. Η συζήτηση όμως πρέπει να συνεχιστεί και όλοι γνωρίζουμε τα αδιέξοδα και τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις μας. Τώρα, έρχομαι στο θέμα της διασφάλισης της προβολής της δράσης μας. Ευχαριστώ πράγματι. Η κατάλληλη προβολή είναι κάτι πολύ σημαντικό για να δείξουμε και στους δικούς μας τους πολίτες την καλή δουλειά που κάνουμε και την στήριξη που προσφέρουμε και να το μάθουν και οι πολίτες των ενδιαφερόμενων χωρών. Εδώ όμως θέλω να μεταφέρω χωριστά την απάντησή μου. Πρώτον, για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, όπου τις μοιραζόμαστε με τον ΟΗΕ. Η ευρωπαϊκή πτυχή, λοιπόν, προβάλλεται όπως οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή επιχείρηση. Και όταν ε, μιλάμε για την προβολή των χωρών μελών, την ε, συμβολή των χωρών μελών δηλαδή στον ΟΗΕ, πρόκειται για εθνική συμβολή. Συνεπώς εδώ ο ΟΗΕ θα έπρεπε να απαντήσει και οι χώρες μέλη. Ε, ζητώ συγγνώμη, αλλά εγώ δεν ξέρω το θέμα αυτό της προβολής πώς διασφαλίζεται στις επιχειρήσεις του ΟΗΕ. Ρωτήσατε κάτι και για τις επιχειρήσεις γεφυρώματος, πώς γίνεται ο σχεδιασμός κλπ. Εδώ, πώς να το θέσω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει τις δυνάμεις της ε, ταχύτατα, παρόλο που πιστεύουμε ότι το κάνουμε αργά, σε σύγκριση με τον ΟΗΕ, αν μη τι άλλο. Οπότε, Στη συζήτηση αυτή που κάνουμε με τους συναδέλφους του ΟΗΕ για το πώς να συνεργαστούμε στην πράξη και πώς να αναπτύξουμε τις κατάλληλες διαδικασίες ώστε αν ο ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει μία επιχείρηση διατήρησης της ειρήνης, πώς αυτό γίνεται στην πράξη. Άρα το θέμα δεν είναι ότι σχεδιάζουμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις ε, με νούμερα στο στάδιο αυτό για στήριξη του ΙΕ. Αυτό που κάνουμε είναι σε διάφορα επίπεδα. Από τη μια ευρύτερη συζήτηση για τις ευρωπαϊκές μάχημες ε, μονάδες, που είναι θέμα του Συμβουλίου και το ξέρετε, αλλά αν αυτό οδηγήσει σε μεγαλύτερη χρήση των ευρωπαϊκών μονάδων, τότε προσωπικά πιστεύω ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό και για συνεργασία με τον ΟΗΕ. Ακόμα όμως δεν είμαστε εκεί. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε πώς και τι και πώς θα μπορούμε να αναπτύσσουμε καλύτερα τέτοιες μάχημες μονάδες ευρωπαϊκές. Τώρα μίλησα για τις διαδικασίες και μπορεί να ακούγεται γραφειοκρατικό, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτοί οι δύο μεγάλοι οργανισμοί να επεξεργάζονται το θέμα της συνεργασίας μεταξύ μας. Γιατί όταν φτάσουμε στη στιγμή να πρέπει να δραστηριοποιηθούμε, δεν έχουμε αυτό το χρόνο. Αυτά πρέπει να έχουν γίνει από πριν. Η Ανίκη συνάδελφος είπε ήδη ότι θα έχουμε ασκήσεις για να ακριβώς δοκιμάσουμε αυτή την ικανότητά μας συνεργασίας όσο γίνεται με πιο γρήγορη αντίδραση. Για τα νούμερα τώρα των Ευρωπαίων πολιτών που εμπλέκονται σε επιχειρήσεις. Και εδώ θα στραφώ στη συνάδελφα από τον ΟΗΕ, γιατί Πρόκειται για πολίτες χωρών μελών, προσωπικό από τις χώρες μέλη, γυναίκες και άντρες που συνεισφέρουν στις επιχειρήσεις του ΟΗΕ. Αλλά από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπαθούμε να προσφέρουμε πλατφόρμες, ευκαιρίες, ώστε ο ΙΕ να μπορεί να απευθύνεται στις χώρες μέλη όταν δεν έχουν αρκετή ικανότητα. Για παράδειγμα, ο κύριος Λατσούς ήρθε στην άτυπη συνάντηση Υπουργών Άμυνα στην Πρατισλάβα πέρυσι και εκεί υποφελήθηκε από την ευκαιρία αυτή και απευθύνθηκε στις χώρες μέλη σε σχέση με τα κενά στην ικανότητα του ΟΗΕ στο Μαλί. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε επαφές με τους συναδέρφους από τον ΟΗΕ για να διευκολύνουμε την συνεργασία με τις χώρες μέλη. Και θέλω από εδώ να ευχαριστήσω για την τόσο καλή συνεργασία που έχουμε με την υπηρεσία του ΟΗΕ εδώ στις Βρυξέλλες, κάτι το οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ για τη συνεργασία αυτή. Συγγνώμη αν δεν τα κάλυψα όλα, θα υπάρξει και δεύτερος γύρος όπως είπατε. Θα επανέλθω λοιπόν. Ευχαριστούμε. Εσείς παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις και νομίζω ότι ε, αφορούσαν το επίκεντρο αυτών που είπα για την ανάγκη μεταρρυθμίσεων στον τομέα της ασφάλειας και της ε, άμυνας. Για το τελευταίο στοιχείο, ε, για το τελευταίο ερώτημα, το... οι 5.549 άνθρωποι αυτοί θα δραστηριοποιούνται ε, υπό τις εντολές του ΟΗΕ και αποτελεί πραγματικά έναν πολύ σημαντικό εταίρο η Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτή την άποψη. Είναι σημαντικό αυτό διότι υπάρχει μια ανισορροπία στον ΟΗΕ. Ε, υπάρχει το Συμβούλιο Ασφαλείας το οποίο δίνει εντολή για συγκεκριμένες επιχειρήσεις και συνέχεια έχουμε ε, υπηκόους Μπαγκλαντές, Νιγηρίας, Ινδίας που εφαρμόζουν αυτές τις εντολές οι οποίες είναι ολοένα και πιο επικίνδυνες. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ε, ε, εκτελούμε αυτές τις πολύ περίπλοκες πλέον επιχειρήσεις. Είναι σημαντικό λοιπόν και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αυξήσουν τη συμβουλή τους και γι' αυτό είναι τόσο θετικό το γεγονός ότι έχουμε αυτήν την ε, πλατφόρμα σε, στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη στη Νέα Υόρκη είναι η, έννοια του TCC, Two Contributing Countries. Troop Contributing Countries, δηλαδή οι χώρες που συνεισφέρουν με στρατηγικές μονάδες ε, που θα, μπορέσει, ε, που θα μας βοηθήσει να υπάρχει ένας καλύτερος σχεδιασμός και συντονισμός για τις μελλοντικές μας επιχειρήσεις. Από πού να ξεκινήσω τώρα για τις ε, αποστολές γεφύρωσης. Ακούστηκαν πολλά. Πράγματι, μιλάμε για μια σχετική ταχύτητα. Φυσικά η, Αφρική, η Αφρικανική Ένωση ε, είχε και εκείνη την ε, συμβολή της. Υπήρχε λοιπόν μια αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης και υπήρχε και η αντίστοιχη αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Παγκή με 350 άτομα για τη σταθεροποίηση της κατάστασης η οποία οδήγησε και στη διάσωση πολλών ανθρώπων και το, η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέδειξε μεγάλη ευελιξία ως προς την ε, διάρκεια αυτής της εντολής προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ε, είχαμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε τις δυνάμεις μας και να προστατεύσουμε τους αμάχους. Αναφερθήκατε επίσης στην, ε, στο Africa Peace Facility. Στη δική σου επιτροπή έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα. Υπάρχει και η πρωτοβουλία Καμπαρούκα, σίγουρα την έχετε ακούσει. Τα κράτη της Αφρικανικής ε, Ένωσης έχουν ε, δεσμευτεί για την αύξηση των, της χρηματοδοτικής συμβουλής έως το 2020 και υπάρχει μια συζήτηση μεταξύ των μελών των, ε, του Συμβουλίου Ασφαλείας ε, για το αν θα μπορούσε ε, να καλυφθεί το 75% του κόστου των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Φυσικά χρειάζεται και λογοδοσία και συγκεκριμένοι μηχανισμοί για να γίνουν όλα αυτά, αλλά είναι σημαντικό ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζήτηση. Η Samantha Power, είχε βοηθήσει πολύ με την ιδιότητά της ε, ως ε, πρέσβυρας. Ε, θα δούμε από εδώ και πέρα πώς θα, πώς προχωρήσει το, η υπόθεση αυτή. Για την προβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ορατότητά της, είναι πράγματι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Κύριε Γκάλερ, αυτό που αναφέρατε, γνωρίζουμε πολύ καλά και εμείς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναγνωρίζεται για την της συμβολή της Τούτου λεχθέντους όμως, όπως είπατε κι εσείς, ε, σε ορισμένες περιπτώσεις ε, τα πράγματα είναι πολύ λεπτά και ευαίσθητα από πολιτικής άποψης και γι' αυτό ενδεχομένως είναι και προς όφελος της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της αλληλοδιαπλοκής των εξωτερικών και εσωτερικών διαστάσεων των ε, εκάστοτε υποθέσεων. Ενδεχομένως λοιπόν ε, κάποιες φορές είναι καλό να βρίσκεται στο παρασκήνιο η Ευρωπαϊκή Ένωση και να προβάλλεται περισσότερο η, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ε, για αυτό αποβαίνει και προς όφελος της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει και μπορεί, να, μπορεί και πρέπει να είναι περήφανη για την συμβολή της στη σταθεροποίηση και στη διατήρηση της ειρήνης στον κόσμο και αυτό μπορεί να ε, χρησιμοποιείται και βεβαίως ως πολιτικό επιχείρημα. Αυτό όμως εμ, ε, πρέπει να σας πω είναι ότι κάποιες φορές είναι καλό να έχουμε τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάποιες φορές είναι καλύτερο να έχουμε τη σημαία του ΟΗΕ. Κάθε φορά, κατά αναπερίπτωση πρέπει να αποφασίζεται το ποιος θα πρέπει να τίθεται επικεφαλής τουλάχιστον ως προς την προβολή και την ορατότητα. Τέλος. Κύριε Νάντ. θέσατε ορισμένα σημαντικά θέματα που μας απασχολούν και μας. Γνωρίζουμε ότι οι πολίτες ανησυχούν και είναι δυσαρεστημένοι με τις αποτυχίες μας. Γνωρίζω πολύ καλά γνωρίζετε κι εσείς το γεγονός αυτό. Ωστόσο, μας ενθαρρύνει το γεγονός ότι σημειώνονται κάποια μικρά ε, βήματα στην πολιτική διαδικασία στο Μαλί που ε, είναι και το επίκεντρο του, του ε, προβλήματος άλλωστε. Χθες εκδόθηκε μια ανακοίνωση ΟΗΕ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, κοινή ανακοίνωση, κάτι που είναι σχετικά συνήθιστο με την οποία ε, χαιρετίζεται η πρόοδος που έχει σημειωθεί. Βεβαίως το, η έκταση της βίας και ο αριθμός των νεκρών είναι ε, πέραν οποιοδήποτε από του ορίου. Έχετε δίκιο σε αυτό και θα πρέπει γρήγορα να αναλυθούν βήματα για να βελτιωθεί η κατάσταση στο, μαλή Στο Και από αυτή την άποψη είναι σημαντικό να ενισχυθεί η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, οι επιχειρήσεις, καθώς και ο αριθμός των εκπαιδευομένων ε, στρατιωτικών. Δεν έχω συγκεκριμένους ε, αριθμούς αυτή τη στιγμή για το ποιος ε, και πόσοι είναι εκείνοι που έχουν αναπτυχθεί, τα μέλη των μονάδων των στρατιωτικών που έχουν αναπτυχθεί, αλλά δέχομαι αυτό που μου λέτε. Και αυτός είναι πράγματι ένας ε, λόγος για τον οποίο απαιτείται ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή και συμμετοχή τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούν τα Ηνωμένα Έθνη μόνα τους να διεκπαιρεώσουν αυτό το καθήκον. Γι' αυτό και χρειάζεται να ενισχυθεί ε, η συνεργασία με τις περιφερειακές ενώσεις, την Αφροκανική Ένωση για παράδειγμα, το G5, ε, που επίσης έχει πάρει σημαντικές πρωτοβολίες και γι' αυτό τον λόγο παροτρύνουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση να διπλασιάσει τις προσπάθειες που καταβάλει. Γιατί η Δυτική Σαχάρα πράγματι εκρεμεί το δημοψήφισμα και εδώ υπάρχει μια πολιτική διαδικασία και υπάρχει και μια επιχείρηση διατήρησης της ειρήνης, επιτόπια. Και εδώ είναι ένα πολιτικό ζήτημα το οποίο πρέπει πρώτα να λυθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει. Μαζί βεβαίως και εκ με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστήσουμε και τις δύο μιλήτριες. Ας περάσουμε τώρα στο δεύτερο γύρο ομιλητών. Θα είναι πιο σύντομος όμως αυτή τη φορά. Έχουμε έναν ομιλητή μόνο, τον κύριο Σαφόιζερ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Όσον αφορά τα ζητήματα ασφάλειας και ανάπτυξης, είχα ασχοληθεί με τα ζητήματα αυτά στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μου και μάλιστα πήγα και στο Καμερούν πρόσφατα για να μελετήσω μαζί με τη βοήθεια των στρατιωτικών πώς έχει η κατάσταση εκεί και με τη βοήθεια κάποιων άλλων κρατών που είναι παρόντα θα ήθελα να δω πώς έχει κατάσταση στη χώρα αυτή και γύρω από τη λίμνη Τσάντ. Συμφωνώ με τα όσα είπε ο Νάρτα όντως υπάρχει ένα πρόβλημα αποτελεσματικότητας. Δεύτερον, τίθεται το εξής ερώτημα. Για ποιο λόγο να αποσυνδέσουμε εντελώ το ζήτημα της ανάπτυξης και το ζήτημα της ασφάλειας στα πλαίσια της χρηματοδότησης. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να έχουμε ασφάλεια χωρίς ανάπτυξη, δεν μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη από την άλλη χωρίς ασφάλεια. Συνεπώς, πρότεινα μια συγκεκριμένη δράση, την οποία θα μπορούσαν να λάβουν στρατιωτικοί, ομοιόμορφες μονάδες μάχης, παντού στην Αφρική, κινητές μονάδες μάχης δηλαδή, οι οποίες θα μπορούσαν να εργαστούν στα πλαίσια μιας επιχείρησης ασφάλειας και ανάπτυξης η Επιτροπή λοιπόν πρέπει να δει πώς μπορεί να χρηματοδοτήσει και τα δύο και πώς μπορεί η ασφάλεια και η ανάπτυξη να μπορούν να κινηθούν μαζί και να φέρουμε και στη χρηματοδότηση όπλων. Αυτό κάποιους ενδεχομένως να τους σοκάρει, αλλά θα πρέπει να δούμε την πραγματικότητα ως έχει. Τρίτον, τίθεται το ζήτημα που έθεσε και ο συνάδελφος Νάρτ πριν από λίγο, το ζήτημα της αποτελεσματικότητας. Δεν πρέπει να δημιουργήσουμε νέους μηχανισμούς. Θα πρέπει να βασιστούμε στην αρχή της επικουρικότητας. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά ποιος είναι παρόν και ποιος δεν είναι παρόν στην Αφρική και ποιος μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά επί Έχουμε τη Γαλλία, τη Ρωσία, στη Βόρεια Αφρική κυρίως, Δεν νομίζω ότι η Γαλλία θα μπορέσει μόνη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα τη Αλγερία, όπου μπορεί να έχουμε πρόβλημα. Το ζήτημα τη Λιβύης επίσης τίθεται, είναι ιδιαίτερα επίκαιρο και εκεί δραστηριοποιείται πάλι ιδιαίτερα η Ρωσία, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό. Συνεπώ έχουμε τη Γαλλία, τη Ρωσία, τι Ηνωμένε Πολιτείε. Είχαμε μια προσέγγιση λοιπόν με τρει παράγοντε. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να ακολουθήσουμε, να δούμε ποιοι είναι σε επιχειρησιακή φάση επιτόπου ποιοι μπορεί να είναι αποτελεσματικοί όχι μόνο για τη διατήρηση της ειρήνης, αλλά θα πρέπει να μπορούν να σκίσουν πίεση, να μπορούν πραγματικά να επιτεθούν αν χρειαστεί, να περιορίσουν ουσιαστικά τις διενέξεις. Νομίζω ότι αυτό πραγματικά θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, θα θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί και νομίζω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουν περισσότερο τους πόλους του G5 Σαχέλ. Μίλησα με τους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είδα επιτόπου, μίλησα επίσης με τους στρατιωτικούς, όλα αυτά σε άτυπο βέβαια επίπεδο. Και μου είπαν, κοιτάξτε, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Συμφωνώ, ωραία, αλλά αν ακολουθήσουμε τις διαδικασίες, τότε πάντα θα είμαστε καθυστερημένοι, πάντα θα υπολοιπόμεθα δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους που ήδη διαθέτουμε, ακριβώς επειδή μας εμποδίζουν συγκεκριμένε διαδικασίες. Μήπως θα έπρεπε λοιπόν να προσαρμοστούμε περισσότερο στην πραγματικότητα. Οι Αμερικάνοι, για παράδειγμα, μας λένε να εργαστούμε με διαφορετικό τρόπο, να έχουμε ένα ταμείο, ένα ταμείο Marshall, το οποίο θα μπορούσε να μας επιτρέψει να χρηματοδοτήσουμε και τις ε, επιχειρήσεις ανάπτυξης αλλά και τις επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης. Μήπως θα έπρεπε λοιπόν να προσαρμοστούμε λίγο περισσότερο στην πραγματικότητα ή θα συνεχίσουμε να φανταζόμαστε επαόριστον ότι κάποια στιγμή η πραγματικότητα θα προσαρμοστεί στις δικές μας διαδικασίες. Και ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να θεωρήσουμε λίγο τη στάση μας. Αυτά που διακυβεύονται είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αν εκραγεί η Αφρική θα εκραγεί και ολόκληρη η Ευρώπη και αυτό ακριβώς βλέπουμε να γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αφρική αν συνεχίσουμε να εργαζόμαστε όπως εργαζόμαστε αυτή τη στιγμή, πραγματικά θα εκραγεί η Αφρική. Δηλαδή η κατάσταση θα βρεθεί εκτός ελέγχου. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν οι ομιλήτριές μας θέλουν να πάρουν το λόγο για να απαντήσουν. Ναι, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον αξιότιμο Ευρωβουλευτή για το ερώτημα το οποίο έθεσε όσον αφορά τη διασύνδεση ασφάλειας και ανάπτυξης. Προφανώς είναι θεμελιώδου σημασία και όλοι συμφωνούν με αυτό. Όντως, θα πρέπει να δούμε πολύ προσεκτικά πώς έχουν οι διαδικασίες μας και πώς μπορούμε να τις βελτιώσουμε. Και όντως, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί έχουμε την σφαιρική στρατηγική πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου πραγματικά εκεί λέμε ότι θα πρέπει να συνεργαζόμαστε περισσότερο με του εταίρου, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, να καταφέρουμε να βελτιώσουμε τι πρακτικέ μα στην Αφρική και το καθεξή. Η σφαιρική λοιπόν στρατηγική πλέον είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχουμε επίση και την ε, Σύνοδο Αφρικής Ένωση, ε, συγγνώμη, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρική που θα λάβει χώρα το φθινόπωρο, στα πλαίσια της οποίας μπορούμε πάλι να εξετάσουμε εκ του σύνεγγυς όλες αυτές τις πτυχές που θίξατε. Και να τονίσω και ένα πιο συγκεκριμένο ζήτημα, έναν τομέα μάλλον όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΕΕ Έθνη έχουν συνεργαστεί και αναφέρομαι στο ζήτημα της διεξαγωγής των επιχειρήσεων και της πειθαρχία. Ξέρετε ότι έχουμε μηδενική ανοχή όσον αφορά τη σεξουαλική κακοποίηση και κατάχρηση. Στον τομέα αυτό έχουμε μία κοινή ανταλλαγή εμπειριών, προτύπων και βέλτιστων πρακτικών με τα Ηνωμένα Έθνη και το λαμβάνουμε αυτό υπόψη μας στην εργασία που κάνουμε αυτή τη στιγμή προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα πρότυπα συμπεριφορά μα. Σα ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι και εγώ εξίσου σύντομη. Συμφωνώ 100% με αυτό που είπατε, διασύνδεση ασφάλεια και ανάπτυξη. Ο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών έχει πει ότι μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε μια βιώσιμη ειρήνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί συγκεκριμένου συμβούλου ειρήνης και ανάπτυξης, προκειμένου να διασυνδεθούν περισσότερα τα πολιτικά θέματα και τα θέματα ανάπτυξης σε χώρες όπου δεν έχουμε αποστολές, όπου δεν έχουμε επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης. Ευχαριστούμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υποστήριξή της αυτήν. Και όντω έχετε απόλυτο δίκιο όταν λέτε ότι είναι το ότι έχουμε πάρα πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες από χώρες όπως η Γαλλία για την καταπολέμηση τρομοκρατίας, για παράδειγμα, στο Μαλί. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα σημαντικότατο παράδειγμα και είχαμε πολύ καλή συνεργασία και με τη Μινούσμα. Καθότι συζητάμε την κεντροφρικανική επίσης δημοκρατία και την κατάστασή της, είναι πολύ σημαντικό να δούμε τις εξελίξεις στη χώρα αυτή και είχαμε μια πολύ επιτυχή συνεδρία δωρητών στις Βρυξέλλες, όπου καταφέραμε να κινητοποιήσουμε περίπου 2 δισεκατομμύρια υπόσχεση τουλάχιστον χρηματοδότησης του ύψου των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό συμβάλλει πάρα πολύ στην παρουσία που έχουμε για τη διατήρηση της ειρήνης στη χώρα αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για τις απαντήσεις σας. Νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε έτσι το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη στο σημείο 5. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Εκτιμούμε όλους ιδιαίτερους την παρουσία σας εδώ. Eh, Θα συνεχίσουμε με το σημείο 6 στην ημερήσια διάταξη. Καλώς. Το τελευταίο λοιπόν σημείο ουσίας τώρα που έχουμε στην εμείς διάταξη είναι το σημείο 6. Αποστολές και επιχειρήσεις της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Αξιοποιούνται τα διδάγματα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Τζοβάνι Κρεμονίνη. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Καλώς ήρθατε. είναι πρόεδρος της ομάδας εργασίας ε, της ΕΚΠΑ για τα, την αξιοποίηση των διδαγμάτων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, το θέμα είναι από τις αποστολές και τις επιχειρήσεις της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Αντιλούμε διδάγματα, τα αξιοποιούμε. Ναι, υπάρχει ένα σύστημα που ισχύει για την αξιοποίηση των διδαγμάτων στα πλαίσια των αποστολών και επιχειρήσεων τη κοινή πολιτική Ασφάλειας και άμυνα. Βέβαια υπάρχουν και περιορισμοί στο σύστημα. Δεν το αρνούμε, δεν πρόκειται για ένα τέλειο σύστημα. Στην παρουσίασή μου λοιπόν, εφόσον μου το επιτρέπετε, θα σας περιγράψω το σύστημα, πώς αυτό λειτουργεί δηλαδή πρώτα απ' όλα. Στη συνέχεια θα διατυπώσω ποια είναι τα όρια και ποια είναι τα πλονεκτήματα του συστήματος που ακολουθούμε σήμερα για την αξιοποίηση διδαγμάτων. Και τέλος θα χρησιμοποιήσω κάποια παραδείγματα διδαγμάτων που πήραμε ή που δεν καταφέραμε να πάρουμε ακόμα. Πρώτον λοιπόν, ποιο είναι το σύστημα που έχουμε στη διάθεσή μας στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για την αξιοποίηση διδαγμάτων. Το σύστημα λοιπόν βασίζεται στο σύστημα του ΝΑΤΟ για τα διδάγματα. Αρχίζουμε λοιπόν με την παρατήρηση των διδαγμάτων αυτών. Στη συνέχεια τα αναλύουμε, τα αξιολογούμε και τι γι' αυτό μιλάμε για τον εντοπισμό των διδαγμάτων, αλλά δεν φτάνει ο εντοπισμό δεν φτάνει η άντληση, πρέπει στη συνέχεια να αναλάβουμε και δράση, να τα αξιοποιήσουμε τα διδάγματα αυτά ώστε να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε. Χρειάζεται λοιπόν αμέσως δράση. Και μόνο εφόσον έχει αναλυφθεί αυτή η δράση μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αξιοποιήσει το δίδαγμα. και αξιοποιείται το δίδαγμα εφόσον έχουμε αλλάξει τις διαδικασίες μας, έχουμε αλλάξει τον τρόπο που δουλεύουμε, τον έχουμε βελτιώσει. Σε πολλά επίπεδα μπορεί να αξιοποιηθούν ε, διδάγματα και σε μεμονωμένες επιχειρήσεις και αποστολές, άλλα διδάγματα περνούν από κάποια διαδικασία στο στρατηγείο μας και υπάρχουν και διδάγματα επίσης τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Πρόκειται για στρατιωτικά και μη στρατιωτικά βέβαια. Το σύστημα για τα στρατιωτικά διδάγματα έχει αναπτυχθεί περισσότερο για ιστορικούς λόγους, από την εποχή του ΝΑΤΟ δηλαδή. Έχουμε όμως και στρατιωτικά και μη στρατιωτικά διδάγματα όπως είπαμε, που αξιοποιούνται στα διάφορα τμήματα. Κάποια από αυτά όμως τα διδάγματα δεν μπορεί να αξιοποιηθούν μεμονωμένα σε ένα συγκεκριμένο τμήμα. Γι' αυτό και συζητιούνται αυτά σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στην ομάδα εργασίας διδαγμάτων της ΚΠΑ, όπου εκεί υπάρχουν εκπρόσωποι διαφόρων τμήματων που μαζί συζητούν τα διδάγματα αυτά. Για παράδειγμα, ένα τέτοιο δίδαγμα που δεν αξιοποιείται από ένα μεμονωμένο τμήμα είναι εκείνο της επικοινωνίας στην ασφάλεια. Οι στρατιωτικές δράσεις και επιχειρήσεις πρέπει να επικοινωνούν με το στρατηγείο. Για να υπάρξει βελτίωση όμως χρειάζεται η βοήθεια του τμήματος πληροφορικής. Γι' αυτό και δεν μπορεί το διδάγμα αυτό να αξιοποιηθεί σε ένα τμήμα μεμονωμένα. Αυτά λοιπόν συζητάει η ομάδα εργασίας για τα διδάγματα της ΚΠΑ όπου έχουμε τις διάφορες δομές της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης ε, με το τμήμα της ΚΠΑ και άλλα. Έχουμε και τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. η, οποία είναι παρούσα με διάφορες υπηρεσίες της, με την Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ, την ΕΚΟ, που σε θέματα ΑΚΠΑ. Υπάρχουν ε, διάφορα προγράμματα ανάπτυξης που έχουν σαν στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας. Τα διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα λοιπόν και αυτά έχουν να κάνουν με το δικό μας έργο της ΚΠΑ και έτσι έχουμε και μια διαφορετική προσέγγιση για το τι πρέπει να βελτιωθεί και πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε καλύτερα μαζί. Διακόπτει ο Πρόεδρος. Πρέπει να πάω σε μια άλλη επιτροπή, οπότε την Προεδρία θα την αναλάβει ο συνάδελφος. Έτσι μην με παρεξηγείτε. Μπορείτε να συνεχίσετε. Πρόεδρος, συγγνώμη κυρίε και κύριοι που πρέπει να φύγω, αλλά πρέπει να πάω να ψηφίσω σε μια άλλη επιτροπή. Σας χαιρετώ λοιπόν. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, τα διδάγματα τα σχετικά με την ΕΚΠΑ και η ομάδα εργασίας για τα διδάγματα της είναι ένα μεγάλο σώμα, έτσι. Είπαμε ότι υπάρχουν θέματα ανάπτυξης, ασφάλειας και είναι καλό που υπάρχει συνεργασία αυτή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί έχουμε έτσι και μια διαφορετική οπτική γωνία. Η συνεργασία μας είναι πολύ καλή για τη βελτίωση του έργου μας. Και όσον αφορά την ασφάλεια και όσον αφορά την ανάπτυξη, μια που εξετάζουμε και τα δύο. Λοιπόν, τι κάνει στην πράξη αυτή η ομάδα εργασία. Με αναφέρθηκα στην άντληση διδαγμάτων πρώτα απ' όλα, τον εντοπισμό του. Συζητάμε ποια είναι τα πιο σημαντικά διδάγματα και ποιε πρέπει να είναι οι προτεραιότητέ μα για την αξιοποίησή τους. Καταλήγουμε λοιπόν κάθε χρόνο σε πέντε διδάγματα κλειδί που εγκρίνονται από τα ανώτατα επίπεδα και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και την Κομισιόν και παρουσιάζεται στη συνέχεια στις χώρες μέλη στην Πολιτική Επιτροπή που τα συζητούν μεταξύ τους. Στη συνέχεια, τρεις φορές το χρόνο συναντιόμαστε με την ομάδα διαχείρισης των διδαγμάτων γιατί είπαμε ότι δεν φτάνει να αντλήσει κανείς τα διδάγματα, να τα εντοπίσει, πρέπει και να τα αξιοποιήσει. Για να σας ε, εξηγήσω τη διαδικασία, τα διδάγματα παραμένουν ανοιχτά μέχρι ότου είτε να υπάρξει αξιοποίησή τους, είτε μέχρι να διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν κάποια αντικειμενικά εμπόδια και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μπορεί να αποφασίσουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο για ένα δίδαγμα, τότε κλείνει. Ποια είναι τα όρια τώρα του συστήματος. Ίσως το έχετε ήδη καταλάβει ότι πρόκειται για ένα εσωτερικό σύστημα. Άρα οι πληροφορίες που έχουμε έρχονται από το εσωτερικό για τα διδάγματα. Βέβαια είναι ένα σύστημα από κάτω προς τα πάνω. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι εργάζονται στην κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας είναι αυτοί οι οποίοι σημειώνουν και λένε στη συνέχεια ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και προτείνουν τι πρέπει να γίνει για να βελτιωθεί. Υπάρχουν διδάγματα βέβαια από σφάλματα τα οποία γίνονται. Και επειδή είμαστε άνθρωποι, πολλέ φορέ δεν θέλουμε να παραδεχτούμε ότι έχουν γίνει σφάλματα. Άρα λοιπόν η αξιολόγηση αυτή δεν θα έλεγα ότι είναι αντικειμενική. Δεν πρόκειται καν για αξιολόγηση. Την αξιολόγηση την κάνει κάποιο που έρχεται απ' έξω. Τα διδάγματα είναι αυτό που έρχεται από μέσα. Και γι' αυτό και υπάρχουν και όρια. Γιατί μερικά διδάγματα μπορεί να μην καταγραφούν καν ή να περάσουν ε, από φίλτρα από την ιεραρχία. Γιατί περνάνε από την ιεραρχία τα διδάγματα. Μπορεί να υπάρξει λογοκρισία επίσης. Και μπορεί να υπάρχουν και διάφορες ε, εκδοχές ενός προβλήματος, οπότε τελικά πρέπει όλοι να αποφασίσουμε ποιο είναι το πρόβλημα πρώτα απ' όλα. Παρά τις δυσκολίες αυτές και τους περιορισμούς, καταφέρουμε να συμφωνήσουμε για διάφορα διδάγματα κλειδί και το πλεονέκτημα του συστήματος αυτού είναι ότι αυτοί οι οποίοι εντοπίζουν τα προβλήματα και τα διδάγματα δεσμεύονται να δουλέψουν πάνω σε αυτά και να τα αξιοποιήσουν κατάλληλα. Γιατί είναι αυτοί που γνωρίζουν καλύτερα την κατάσταση, αυτοί κάνουν τη δουλειά επιτόπου και έτσι υπάρχει μια ανάλυση στην οποία συμμετέχουν ε, όλα τα μέλη της ομάδας εργασίας για το πώς θα προχωρήσουμε στη συνέχεια. Υπάρχει λοιπόν αυτή η δέσμευση για πρόοδο και υπάρχει και μια πίεση μεταξύ ομοτήμων ότι δηλαδή πρέπει να παρουσιάσουμε την πρόοδο που έχουμε επιτύχει. Πώς αξιοποίησαμε δηλαδή τα διδάγματα αυτά. Είναι και αυτό κίνητρο για να προχωρήσει κανείς και να βελτιώσει τη δουλειά του. Θα σας δώσω τώρα μερικά παραδείγματα διδαγμάτων κλειδί που εντοπίσαμε τα τελευταία χρόνια. Ένα που έχω στο μυαλό μου είναι το γεγονός ότι χρειάζεται κατάρτιση πριν το στάδιο ανάπτυξης για όλο το προσωπικό που συμμετέχει σε επιχειρήσεις και αποστολές. Μπορεί να φαίνεται αυτό προφανές, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχει περάσει από την κατάρτιση αυτή ολόκληρο το προσωπικό πριν συμμετάσχει σε μια αποστολή ή δράση. Οι χώρες μέλη προσφέρουν κατάρτιση, όχι όλες, άλλες ναι, άλλες όχι, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο για όλο το προσωπικό. να μαθαίνει δηλαδή ο κόσμος που συμμετέχει σε αυτές, τι ακριβώς είναι αυτές οι αποστολές, ε, οι αντιπροσωπείς Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, ποιες είναι οι βέλτιστες ε. πρακτικές. Έχουμε τέτοια σεμινάρια λοιπόν κάθε μήνα εδώ στις Βρυξέλλες που γίνονται σεμινάρια κατάρτισης που γίνονται σε θελοντική βάση όμως, όχι υποχρεωτικά. Οπότε το επόμενο στάδιο είναι να γίνουν υποχρεωτικά για όλο το προσωπικό μας. Θα συμπεριλαμβάνεται αυτό στη νέα πολιτική κατάρτιση της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Βλέπετε, έτσι δουλεύουν τα πράγματα, έτσι μετά τον εντοπισμό έχουμε τις συστάσει και μετά έχουμε την υλοποίηση. Ένα άλλο δίδαγμα είναι το θέμα της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ ε, αποστολών ΟΚΠΑ με την Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ έχουμε συγκεντρώσει κάποιες βέλτιστες πρακτικές από αποστολές και επιχειρήσεις επιτόπου. Συγκεντρώνονται αυτές οι βέλτιστες πρακτικές σε κατευθυντήριες γραμμές. Μπορεί κανείς ε, να σκεφτεί ότι είναι σαφές τι πρέπει να κάνει η αντιπροσωπεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Όμως δεν είναι τόσο προφανές γιατί υπάρχουν και κάποιες γκρίζε ζώνες. Συντονισμό με δωρητέ με την χώρα υποδοχή, Οι κατευθυντήριε αυτές γραμμές λοιπόν βέλτιστων πρακτικών μας καθοδηγούν κάπως για το τι να κάνουμε για να συνεργαστούμε καλύτερα, να αποφύγουμε τις επικαλύψεις επιτόπου μεταξύ της EUSR, των ε, αντιπροσωπιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αποστολών επιχειρήσεων ΚΠΑ. Και ένα άλλο παράδειγμα, δίδαγμα το οποίο δεν αξιοποιήθηκε, έχει να κάνει με τις ασφαλείς επικοινωνίες. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν έχουμε σύστημα ασφαλών επικοινωνιών ανάμεσα το στρατηγείο μας στις Βρυξέλλες και τις διάφορες ε, ε, αποστολές και επιχειρήσεις. Δεν έχουμε ε, ασφαλή τηλεφωνική επικοινωνία. Οπότε χρησιμοποιούν τα εθνικά συστήματα ασφάλειας της πρωτεύουσας, στη χώρα αποδοχής που βρίσκονται, με το στρατηγείο μας αλλά ούτε καν στι Βρυξέλλε με τα διάφορα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν έχουμε ασφαλεί επικοινωνίε Είναι κάτι που μας λείπει. Υπάρχουν διαφορετικά συστήματα που δεν επικοινωνούν μεταξύ του. και αυτό είναι πρόβλημα. Παραμένει λοιπόν ένα ανοιχτό δίδαγμα και θα παραμείνει ανοιχτό γιατί ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι, να αξιοποιήσουμε και αυτό το δίδαγμα. Γι' αυτό και παραμένει. Συνεπώ. συμπερασματικά, ελπίζω ότι σας έπεισα πως έχουμε ένα σύστημα για την αξιοποίηση διδαγμάτων. Βέβαια το σύστημα δεν είναι τέλειο. Έχει περιορισμούς, έχει όμως και πλεονεκτήματα. Κατά τη γνώμη μου υπάρχει θετική τάση όσον αφορά την αξιοποίηση των διδαγμάτων. Τη δουλειά αυτή την κάνω εδώ και αρκετά χρόνια και πιστεύω ότι οι επιχειρήσει και αποστολέ γίνονται πιο επαγγελματικέ, πιο αποτελεσματικέ ή βέβαια μια διαδικασία που προχωράει αργά. Αλλά Είναι βέβαια μια διαδικασία που προχωράει αργά, αλλά η τάση είναι προ τη βελτίωση. Σημειώνω επίση και την καλή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ των υπηρεσιών στην ομάδα εργασία διδαγμάτων, για παράδειγμα, όπου εντοπίζονται και αξιοποιούνται στη συνέχεια τα διδάγματα. Υπάρχει συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να λάβουμε υπόψη μας και την διάσταση της ασφάλειας και την διάσταση της ανάπτυξης. Και σας διαβεβαιώ ότι στην ομάδα εργασίας διδαγμάτων της ΚΠΑ θα συνεχίζουμε να δούμε διδάγματα μαζί και θα συνεχίσουμε να προωθούμε και να ελέγχουμε και την αξιοποίησή τους. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κύριε Κρεμονίνη. Πρωτού δώσω το λόγο στις πολιτικές ομάδες, θα ήθελα να θέσω εγώ ένα ε, ερώτημα. Πρώτον, αξιοποίηση δαγμάτων Δεδομένου του ότι σε τελική ανάλυση η μορφή αποφασίζεται από την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας. Μας δώσατε ένα παράδειγμα για ένα δίδαγμα που δεν είχε αξιοποιηθεί επαρκώς. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, οι προτάσεις σας ε, λαμβάνονται υπόψη ή απλώς ε, γίνονται αντιληπτές ως ε, διοικητική συμβουλή. Για τις κρατικές προμήθειες σε σχέση με τις αποστολές, τις αναπτυξιακές επιχειρήσεις που κάναμε για παράδειγμα στη Γεωργία, χρειάστηκαν έξι μήνες για να προκυρηθεί διαγωνισμός για, τη, για τα καύσιμα. Χρειάστηκαν έξι μήνες λοιπόν έως ότου καταφέρει η αποστολή να αποκτήσει επιχειρησιακή ικανότητα λόγω του ότι δεν γινόταν ο διαγωνισμός για τα καύσιμα. Οπότε το ερώτημά μου είναι τι πιστεύετε, ε, σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι έχει αλλάξει η φύση των αποστολών. Και δεύτερον, δεν υπάρχει ένα σύστημα κεντρικής έκδοσης εντολών. Εσείς προτείνετε να ε, ε, να υπάρξει κάποιος εκ των προτέρων σχεδιασμός ή προτείνεται να έρχεστε εκ των υστέρων μετά τις αποστολές να κάνετε κάποιες, ε, έναν απολογισμό και κάποιες αντίστοιχες προτάσεις ή θέλετε κι εσείς ή αντιθέτως ε, ε προτείνεται να δημιουργηθεί ένα κέντρο σχεδιασμού. Ο κύριος Γκάλερ. Ευχαριστώ πολύ. Αν μιλάτε γερμανικά, ε, βεβαίω πολύ, πολύ ωραία, δεν χρειάζεται να βάλετε τα ακουστικά σας. Αλλιώς βάλτε τα σας παρακαλώ. Και εγώ θα ήθελα στο πλαίσιο αυτών, αυτής της των διδαγμάτων και των αντιστοίχων διαδικασιών που εφαρμόζεται να προβλέπετε η δυνατότητα να κατανομάζονται τα πράγματα με το όνομά τους. γιατί πολλές φορές έχουμε δει ο λόγος να αμβλύνεται, να προσπαθούμε να, να γίνονται προσπάθειες να ε, εξομαλυθούν ίσως κάποιες ε, γωνίες ως προς τη διατύπωση που χρησιμοποιείται ε, και έτσι πολλές φορές δεν γίνεται και σαφές πού ακριβώς υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης. Επίσης, ως προς τα διδάγματα, εγώ θα διέκρινα δύο σφαίρες. Πρώτον, είναι η σφαίρα εκείνων που μπορούμε να κάνουμε εμείς και δεύτερη η σφαίρα ε, που αφορά την χώρα υποδοχής, την, ε, την χώρα φιλοξενίας. Ε, υπήρχε για παράδειγμα ε, μια δραστηριότητα για την αστυνομία του Κονγκό. Αν όμως ο κύριος Καμπίλα δεν έχει καμία απολύτως πολιτική, πολιτική βούληση να συνδράμει σε κάτι που θα ενίσχυε τη σταθεροποίηση της ίδιας του της χώρας, ε, τότε τι να κάνουμε, ατυχήσαμε. Το ερώτημα λοιπόν που πρέπει να θέτουμε στον εαυτό μας είναι εκ των προτέρων, ακόμη και αν έχουμε λάβει πρόσκληση υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει περίπτωση να βελτιώσουμε ή να επηρεάσουμε θετικά τα πράγματα. Φυσικά καλό είναι να γίνεται και ένας εξπόστα απολογισμός, εκ των υστέρων ε, απολογισμός, αυτό που κάνετε εσείς, αλλά καλό θα ήταν να γίνεται και, ένας, και μια εξάντε αξιολόγηση ε, του ποιες είναι οι δυνατότητες που έχουμε γιατί αν έχει γίνει μια τέτοια αξιολόγηση, είναι και πολύ καλύτερη και πολύ πιο αποτελεσματική η εκπαίδευση που μπορούμε να προσφέρουμε στο προσωπικό μας. Χρειαζόμαστε σε κάποιες περιπτώσεις ε, μαχητές, στρατιωτικούς οι οποίοι θα ρηχτούν στη μάχη. Τώρα το κάνει η Γαλλία ε, στο Μαλί αλλά καλό θα ήταν να αλλάξει η μορφή αυτής της παρέμβασης και να γίνει πιο, πιο ολοκληρωμένη και πιο συνολική. Άλλο ερώτημα. Πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει και να βελτιωθεί η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Προς το παρόν έχουμε το MCCP, το οποίο αφορά την ε, κατάρτιση. Θα βοηθήσει αυτή η διαδικασία ε, της, ε, την δυνατότητα και τις ικανότητες επιχειρησιακής δραστηριοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή θα υπάρξουν πιστεύετε και νέες χρηματοδοτικές δυνατότητες για το μέλλον κάτι που βεβαίως θα επηρεάσει επί και τα διδάγματα που αντλούνται. Ευχαριστώ, έχω δύο ακόμα ομιλητές. Στη συνέχεια προτείνω να δώσουμε το λόγο στον προσκεκλημένο μας ε, και για να μην ξεχαστούν και τα ερωτήματα που τέθηκαν μέχρι στιγμή. Κυρία Χολέρο. Ευχαριστώ πολύ. Δύο σύντομα ερωτήματα έχω να θέσω. Είναι περίεργο το γεγονός ότι δεν έχουμε ακόμη αξιοποιήσει τα διδάγματα για τις επικοινωνίες ασφαλείας. Πώς είναι δυνατόν σήμερα, στη σημερινή εποχή, να μην έχουμε ακόμα καταφέρει ε, να έχουμε ασφαλείς επικοινωνίες. Επίσης, αναρωτιέμαι, έχετε ε, συζητήσει ποτέ το θέμα της ισορροπίας των, των φύλων. Υπάρχουν διδάγματα σε αυτόν τον τομέα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Ε, ο κύριος Σαφχοίζα. Oui, Σε σχέση με το θέμα το οποίο μας απασχόλησε μόλις πριν, να πω κάτι. Εγώ θα ήθελα να γίνει ένας έλεγχος, ένας εξωτερικός έλεγχος. Πρώτον, όσον αφορά πώς μπορούμε να συνδέσουμε περισσότερο την ασφάλεια και την ανάπτυξη για τη χρηματοδότηση, τη διάρθρωση, την οργάνωση. Είναι θεμελιώδου σημασία σε αυτό το ζήτημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διασυνδεθούν και τα δύο αυτά, ασφάλεια και ανάπτυξη, στις δομές και στην οργάνωση και στη χρηματοδότηση βέβαια. Δεύτερον, είχαμε και έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα G5 Σαχέλ, με πολλά δισεκατομμύρια ευρώ για την ασφάλεια και την ανάπτυξη. Για ποιο λόγο δεν λειτουργεί όμως? Για ποιο λόγο δεν βρίσκεται πραγματικά στο ύψος των απαιτήσεών μας επιτόπου. Θα ήταν ενδιαφέρον και αυτόν το διερευνήσετε λίγο. Η αρχική ιδέα είναι πολύ καλή για το πρόγραμμα αυτό, αλλά δεν ανταποκρίνεται στις περιστάσεις και δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες και στις ανάγκες χρηματοδότησης και τις οργανωτικές ανάγκες των επιχειρήσεων. Να λοιπόν κάποιες εμπειρίες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν χρήσιμα διδάγματα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κρεμονίνη, λοιπόν, ακούσατε τις παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις των συναδέλφων. Έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ε, καλές αυτές ερωτήσεις. Πρώτον, διευκρινήσεις όσον αφορά την ακολουθητέα διαδικασία, το ρόλο της ομάδας εργασίας μας και τι συνέχεια δίδεται. Η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας των κρατών μελών μέχρι στιγμής έχει εφαρμόσει όλα αυτά τα κέρια διδάγματα, το σύστημα που σας περιέγραψα άρχισε να λειτουργεί το 2013. Τα βασικά διδάγματα, τα κέρια αυτά διδάγματα ήταν αρκετά γενικά, πρέπει να το παραδεχτώ αυτό και διατυπωμένα με τρόπο διπλωματικό ώστε να γίνουν αποδεκτά από όλα τα κράτη-μέλη, τα οποία διαφορετικά θα τα αρνούνταν. Προφανώς θα πούνε να χρειαζόμαστε ασφαλείς επικοινωνίες. Το πιο σημαντικό είναι να εγκρίνουν καταρχά τα διδάγματα τα κράτη-μέλη, πράγμα το οποίο το έχουν κάνει για τα διδάγματα που έχει προτείνει η ομάδα εργασία μου. Εναπόκειται σε εμά όμω έπειτα να αναλάβουμε δράση προκειμένου να εφαρμοστούν στην πράξη τα διδάγματα αυτά. Την εντολή για την εφαρμογή μα τη δίνουν τα κράτη-μέλη. Πρέπει λοιπόν εμεί να κάνουμε μια συγκεκριμένη εργασία προκειμένου τα διδάγματα να εφαρμοστούν στην πράξη. Προκειμένου λοιπόν να γίνει κάτι τέτοιο, απαιτούνται αρκετέ προσπάθειε από εμά. Όσο και διαμαγεία δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί και πολλέ φορέ η διαδικασία είναι αρκετά χρονοβόρα και αργή. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι σημειώνουμε πρόοδο. Είπατε κι εσεί όντω υπάρχουν προβλήματα με τις δημόσιες προμήθειε. Δεν ξέρω πότε συνέβη το επεισόδιο αυτό με τη βενζίνη που είπατε στην αποστολή της Γεωργίας. Ναι, αλλά πότε σας ρωτάω ποια χρονική περίοδο. Πρόεδρος, η ε, επιχείρηση παρατήρησης αυτή η μεθοριακή ήταν πριν από 3,5 χρόνια. Αποτελέσαμε εμείς ε, μία συνέχιση της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών και έπειτα έγινε μία δημόσια προσφορά για παροχή καυσίμων για 7 μήνες. Κοιτάξτε, η διαδικασία δημοσίων συμβάσεων είναι κάτι το οποίο πρέπει να επεξεργαστούμε περισσότερο. Οι μη στρατοτικέ αποστολές όπως αυτή της Γεωργίας βρίσκεται υπό τη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, μιας συγκεκριμένη διεύθυνση, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αρμόδια για τη χρηματοδότηση και για τι δημόσιες συμβάσει και για τι δημόσιες προμήθειες. Συνεπώς πολλές φορές υπάρχει μια αναντιστοιχία αν θέλετε στη συμμετοχή των δύο αυτών οργάνων, ΕΕΔ και Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όντως κάποια λάθη έχουν γίνει, το αποδεχόμαστε αυτό, δεν είμαστε αποτελεσματικοί εν προκειμένου. Δεν συμβαίνουν όμως τα συμβάντα αυτά τόσο συχνά. Ξέρετε ότι μπορούμε εμεί να κατηγορήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να τη πούμε ότι δεν ήταν αρκετά αποτελεσματική αλλά οι υπηρεσίε Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μα απαντήσουν όχι, το δικό σα δικό σας είναι το λάθο, γιατί εσεί δεν κάνατε έναν πρώτερο σχεδιασμό. Βρήκα όμω τώρα κάποιον τρόπο προκειμένου να συνεργαζόμαστε καλύτερα, να έχουμε μια κοινή συνεργασία δηλαδή αποτελεσματική ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακριβώ ότι συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΕΔ στα πλαίσια τη ομάδα εργασία για τα διδάγματα τη κοινή πολιτική άμυνα και ασφάλεια είναι κάτι το πάρα πολύ θετικό. Το πρόβλημα αυτό πάντως προέκυψε πριν από κάποια χρόνια, έτσι δεν είναι πρόεδρος. Με διαδικασία δημοσίων προμηθειών είναι ήδη, γιατί εσείς δεν δεχτήκατε την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προσαρμοστεί εκ νέου η διαδικασία αυτή. Και έτσι κατά αυτόν τον τρόπο συνεχίζεται η διαδικασία αυτή. Είδαμε με το Ισραήλ μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε προκειμένου να δημιουργηθεί ένας κόμβος προσγείωσης των ελικοπτέρων, δεν, έγινε δεχθή η αρχική πρόταση των Ισραηλινών, χρειάστηκε να περάσουν τρει-τέσσερι μήνε προκειμένου να έχουμε την προσφορά από κάποιο άλλο κράτο. Και στο τέλο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι δεν χρειαζόμαστε ενδεχομένω διαδικασία αυτή. Εγώ νομίζω ότι να λειτουργούμε ad hoc κάθε φορά θα πρέπει να υπάρχει μια θεσμοθετημένη εκ των προτέρων κοινή διαδικασία που να ακολουθείται κάθε φορά. Ο κύριο Κρεμονίνη ναι, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις όντως και από τις διαφορετικές υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν βρίσκομαι εδώ πέρα βέβαια όμως για να ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από όσο ξέρω όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να επιταχύνει λίγο τις διαδικασίες της. Αν υπάρχει παράλληλα και ο κατάλληλος σχεδιασμός θα καταφέρουμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία και για τις δημόσιες προμήθειες. Όντως δεν έχουμε σημειώσει πρόοδο στον τομέα αυτό και όντως αξίζει να διερευνήσουμε περισσότερο αυτά, τα είπατε, αυτά που είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος ε, ε, Σαν Σονχάζερ, να συμφωνήσω με τον πρόεδρο όμω, γιατί τα ίδια προβλήματα έχουμε δει και στην Αφρική, όπου έχουμε πάρα πολύ αργέ διαδικασίε όσον αφορά τι δημόσιε συμβάσει. Ο κύριο Κρεμονίνη Κοιτάξτε, κάθε φορά υπάρχουν κανόνε και πρέπει να ακολουθούμε του κανόνε και βέβαια αυτό πρέπει να γίνεται αποτελεσματικά και γρήγορα. Εκείνη η πρόκληση. Ναι, αλλά ξέρετε ότι οι Αμερικάνοι καταφέρνουν και οργανώνται διαφορετικά όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Το κάνουνε. Για ποιο λόγο και εμεί δεν μπορούμε να μιμηθούμε του Αμερικανού. Πρόεδρο. Κοιτάξτε, για να καταλαβαίνουμε ακριβώς τι κάνουμε και εδώ πέρα, ε, δεν μιλάμε για κάτι το οποίο δεν έχουμε καλύψει ποτέ στο παρελθόν, η δική μας Επιτροπή είχε πει ότι θα έπρεπε να εγκριθούν διαφορετικοί κανόνες όσον αφορά τη χρηματοδότηση και όσον αφορά τις α, δημόσιες προμήθειες. Ότι θα πρέπει και τις δημόσιες προμήθειες να ακολουθούν τη δικασία που ακολουθείται γενικότερα για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Η πρόταση η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απορρίφθηκε, μολονότι εμεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια επιμένουμε πάρα πολύ στην αλλαγή των κανόνων. Δυστυχώ οι κανόνε όμω δεν τροποποιήθηκαν και γι' αυτό το λόγο ακολουθούμε του κανόνε που ακολουθούμε στι δημόσιε προμήθειε. Και ξέρετε ότι πολλέ φορέ δεν καταφέρνουμε να είμαστε πιο ευέλικτοι στι δημόσιε προμήθειε γιατί δεν άλλαξαν οι κανόνε. Εμεί ε, ω Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιμείναμε προκειμένου να αλλάξουν οι κανόνες, αλλά η πρότασή μα στον τριμερή διάλογο απορρίφθηκε. Ο κύριο κρεμονίνη θα μπορούσαμε να εμβαθύνουμε περισσότερο στο ζήτημα αυτό, αν έχουμε μια ειδική συνεδρίαση. Γι' αυτό θα μπορούσαν να έρθουν οι συνάδελφοι από το FPI της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την Υπηρεσία δηλαδή Μέσων εξωτερική πολιτική για να το συστήσουμε περαιτέρω το ζήτημα αυτό. Τώρα, αν η αξιοποίηση των διδαγμάτων όντω έχει αντίκτυπο επιτόπου σε κάποιε επιχειρήσει. Θεωρώ πω ναι. Ξέρετε ότι ε, σαφώς θα πρέπει η άντληση και αξιοποίηση των δαγμάτων να έχει θετικές επιπτώσεις και επιτόπου και έχει θετικές επιπτώσεις στο συντονισμό, στην ασφάλεια Ελπίζω λοιπόν ότι όντω υπάρχει μια άμεση, ένας άμεσος αντίκτυπος θετικός επιτόπου κάθε φορά που αξιοποιούμε και αντλούμε διδάγματα. Ασχολούμεθα μόνο με λεπτομέρειες των επιχειρήσεων ή και με πιο στρατηγικά ζητήματα. Κοιτάξτε, εμείς δεν πάμε τόσο μπροστά, να ταινίζουμε τόσο μακριά το μέλλον. Προσπαθούμε να δούμε λίγο τι είχε συμβεί στο παρελθόν. Αντλούμε διδάγματα αποσφάλματα του παρελθόντος. Βάσει αυτών λοιπόν κάνουμε συγκεκριμένε προτάσεις οι οποίε θα πρέπει όμως να εγκριθούν στη συνέχεια και από την ιεραρχία μας. Δεν μπορούμε εμεί να κάνουμε μια πολύ φιλόδοξη, τολμηρή πρόταση, αν αυτή τελικά μετά δεν εγκριθεί από την ιεραρχία μας δεν θα έχει κανένα αντίκρισμα. Μην περιμένετε εμεί να σα δώσουμε ένα νέο όραμα για τον έλεγχο και τη διοίκηση Εμεί προσπαθούμε να εντοπίσουμε διδάγματα και να κάνουμε συγκεκριμένε συστάσει στη συνέχεια, οι οποίε βέβαια μπορεί κάποια στιγμή να οδηγήσουν και σε κάποιε πρωτοβουλίε στρατηγική φύση. Αλλά επαναλαμβάνω, βασιζόμαστε περισσότερο στην εμπειρία του παρελθόντο και προσπαθούμε να είμαστε συγκεκριμένοι και αντικειμενικοί ω προ το τι πρέπει να γίνει για να αλλάξουν τα συγκεκριμένα προβλήματα. Ο κύριος Γκάλερ στη συνέχεια αναφέρθηκε σε κάποια ζητήματα Όντως, προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο σαφείς και συγκεκριμένοι και διαφανείς γίνεται. Μερικές φορές όμως στη διατύπωση των διδαγμάτων πρέπει να είμαστε και κάπως διπλωματικοί. Διότι καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τον ένα και τον άλλο για τη διάπραξη συγκεκριμένων σφαλμάτων και όλοι τελικά πρέπει στο να συμφωνούμε για τον δρόμο που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Και πολλές φορές όντως η διατύπωση ενδεχομένως να ακούγεται κάπως διπλωματική, αλλά αυτό είναι αναγκαίο τελικά αν θέλει κανείς να συμφωνήσει και όντως να αξιοποιήσει τα διδάγματα. Στη συνέχεια, τα διδάγματα αυτά μπορούν μέσω συγκεκριμένων πια δράσεων να εφαρμοστούν. Αυτές οι δράσεις προφανώς θα πρέπει να είναι σαφείς και συγκεκριμένες. Στη συνέχεια το ζήτημα των χωρών υποδοχής. Πάλι εδώ πέρα δικός μας τρόπος εργασίας επηρεάζει τα πράγματα. Πάντως, εν γέννη προκειμένου μια αποστολή επιχείρηση να είναι αποτελεσματική θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και το τοπικό περιβάλλον, το τι ισχύει επί τόπου. Είπαμε ότι υπήρχε ένα κύριο βασικό δίδαγμα όσον αφορά το local ownership, να υπάρχει δηλαδή ένας ενστερνισμός των αρχών μας από την τοπική κοινωνία, από τη συγκεκριμένη αυτή χώρα στην οποία δραστηριοποιούμεθα. Προκειμένου όμως να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει και εμείς να αναλύσουμε τις συνθήκες που ισχύουν σε μια συγκεκριμένη χώρα να δούμε ακριβώς ποιο είναι το συγκεκριμένο πλαίσιο το οποίο ισχύει στη χώρα αυτή, προτού προχωρήσουμε στο σχεδιασμό μιας επιχείρησης. Και έχουμε και ένα άλλο δίδαγμα, το οποίο λέγεται πολιτικό πλαίσιο όσον αφορά την προσέγγιση συγκεκριμένων κρίσεων, όπου προσπαθούμε μέσω ενό εγχειριδίου ουσιαστικά να έχουμε μια κοινή ανάλυση μεταξύ Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων για το πώ μπορούμε να αναλύουμε συγκεκριμένε περιπτώσει κρίσεων και να δούμε ποια είναι όλα τα εργαλεία τα οποία εμεί έχουμε στη διάθεσή μα εργαλεία από τα οποία πολλές φορές βρίσκονται εκτό κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνας. Και αφού γίνει η ανάλυση αυτή με τα διαθέσιμα εργαλεία, τότε καλούμεθα εμεί να αποφασίσουμε αν αξίζει ή όχι να επέμβουμε επιτόπου και να λάβουμε υπόψη μας επίσης και την τοπική νοοτροπία που υπάρχει σε μια χώρα. Προφανώς και αυτό πρέπει να γίνει. Ορισμένα πράγματα μπορούμε να τα κάνουμε, αλλά πάλι όχι. Αναφερθήκατε στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Υπάρχουν εκεί συγκεκριμένοι περιορισμοί. Συμφωνώ μαζί σας ότι αυτοί θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Προσπαθούμε στην ανάλυση που κάνουμε να αντικατοπτρίζεται και η τοπική κατάσταση και προσπαθούμε αυτό να το κάνουμε βέβαια εκ των προτέρων, προτού ληφθεί συγκεκριμένη απόφαση για την εξαγωγή μια επιχείρησης. Επίσης, η ομάδα εργασίας για τα διδάγματα της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας έχει καταλήξει και σε κάποιες κατευθύνες γραμμές για το πώς μπορεί να συντάξει κανείς ένα πλαίσιο ανάλυσης ε, προτού επέβουμε σε μια συγκεκριμένη περιοχή, δηλαδή προτού στηθεί μια επιχείρηση. Και πρέπει να δούμε και να έχουμε και τις κατάλληλες επιχειρήσεις τελικά. Αναφερθήκατε στο Μαλί, αναφερθήκατε και σε άλλες χώρες κάνουμε και στρατηγικές αναθεωρήσεις, αξιολογήσεις μάλλον, οι οποίες ελπίζω ότι ασχολούνται με το ζήτημα το οποίο θίξατε. Ελπίζω ότι αυτές οι αναθεωρήσεις μας επιτρέπουν να τροποποιήσουμε ακόμα και να σταματήσουμε κάποιες επιχειρήσεις. Αν τα κράτη-μέλη θεωρήσουν ότι για παράδειγμα είναι ανεπαρκής ή ότι δεν προσαρμόζονται στην τοπική κατάσταση. Τώρα, αν με τη νέα ΠΕΣΚΟ τα πράγματα θα βελτιωθούν. Η ΠΕΣΚΟ εφόσον λάβει χώρα, η MPCC θα λάβει χώρα. Εμείς ως ομάδα εργασίας για τα διδάγματα θα πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσουν αυτοί οι δύο φορείς. Θα έχουμε λοιπόν μια νέα δομή, μια νέα διάρθρωση. Προφανώς θα γίνει μια άντληση διδαγμάτων για την εργασία των δύο αυτών δομών και βάσει των διδαγμάτων αυτών φαντάζομαι και εμεί ότι θα καταφέρουμε να προτείνουμε κάποιες διορθωτικές δράσεις ή κάποιες βελτιωτικέ δράσεις. Και αυτό λοιπόν θα μας απασχολήσει. Κύριε Βαλέρο, έθεσε κάποια ζητήματα. Για ποιο λόγο δεν αντλήσατε διδάγματα όσον αφορά τι ασφαλεί επικοινωνίε, Μα προσπαθήσαμε και προσπαθούμε. Έχουμε απόλυτη συνείδηση του προβλήματο, αλλά είναι αρκετά δύσκολα τελικά τα πράγματα. Πέρυσι προσπαθήσαμε να ξεκινήσουμε ένα διαγωνισμό υποβολής προσφορών για ένα νέο σύστημα, το EC3IS, ένα νέο σύστημα ασφαλών επικοινωνιών που θα καλύπτει και έτσι την προσωπία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το κεντρικό μας στρατηγείο. Αλλά η διαδικασία αυτή υποβολής προσφορών απέτυχε γιατί δεν είχαμε την απαραίτητη, τον απαραίτητο προπολογισμό. Λάβαμε κάποιες προσφορές οι οποίες δεν αντιστοιχούσαν τελικά στα ποσά τα οποία εμεί θα μπορούσαμε να δώσουμε. Άρα η διαδικασία ξεκινάει τώρα πάλι από την αρχή. Έχουμε, αν θέλετε, και περιορισμού τέτοια φύση. Περιορισμοί λοιπόν χρηματοδοτικοί, το ότι κάποιε διαδικασίε είναι χρονοβόρε, όλα αυτά δεν βοηθούν, αλλά σαφώ συνειδητοποιούμε ότι είναι προβληματικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να βελτιώσουμε. Γι' αυτό παρακολουθούμε τα ζητήματα αυτά εκ του σύναγγη. Ισορροπία και εκπροσώπηση των δύο φύλων. Και ξέρετε ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη μελέτη που έγινε από τους συναδέλφους της μη στρατιωτική δυνατότητα σχεδιασμού και διεξαγωγής επιχειρήσεων της CPCC, όπου ασχολήθηκαν, αν θέλετε, με την διάσταση της εκπροσώπησης των δύο φύλων, άρα και το ζήτημα αυτό μας απασχολεί. Τέλος. Άλλες πιθανές εμπειρίες όσον αφορά την ανάπτυξη και την ασφάλεια. Κοιτάξτε, στην ομάδα αυτή εργασίας για τα διδάγματα μετέχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΕΔ. Προσπαθούμε να δούμε τη διασύνδεση ανάμεσα στην ανάπτυξη και την ασφάλεια. Αυτό μας ενδιαφέρει κυρίως βέβαια είναι οι αποστολές και επιχειρήσεις της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Δεν θα πάμε δηλαδή να αντλήσουμε διδάγματα από πράγματα τα οποία διαχειρίζεται αποκλειστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορούμε να συγκρίνουμε τη δική μας εργασία με τη δική τους, αλλά εμείς ως ΕΕΔ αναγκαστικά επικεντρωνόμαστε σε αποστολές και επιχειρήσεις της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Αυτές θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη μας το γενικότερο πλαίσιο της διασύνδεσης ασφάλειας και ανάπτυξης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Άλλες ερωτήσεις? Όχι δεν βλέπω. Οπότε, μια που δουλεύουμε και στην διάμεση αναθεώρηση του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου, κάντε ένα κατάλογο για τις προτάσεις που κάνετε και σε τι βαθμό έχουν ληφθεί ήδη υπόψη όχι, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε μια καλή επισκόπηση των διδαγμάτων που αξιοποιήθηκαν και θα ξέρουμε από την Πολιτική Επιτροπή τι έχει αξιοποιηθεί και τι όχι. Από την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας. Γίνεται, είναι εφικτό αυτό. Ναι, βέβαια τα έγγραφα αυτά είναι περιορισμένα. Θα δούμε τους συναδέρφους και ποιοι είναι οι κανονισμοί για το τι μπορούμε να μοιραστούμε μαζί σας ή όχι. Εννοείται, αλλά πάντως αν το επιτρέπουν οι κανόνες θα ήταν πολύ καλό, αλλιώς άτυπα θα έπρεπε να ζητήσουμε μήπως μπορούμε με κάποιο όλο τρόπο να τα πάρουμε. Αν δεν είναι εμπιστευτικά, αν μη τι άλλο, θα μπορέσετε να μας δώσετε μια ιδέα Και όσο προχωράει η κατάσταση, το Κοινοβούλιο πολύ χαίρεται και θέλει να το ξέρει αυτό, πόσο προχωράνε. Λοιπόν, ευχαριστούμε που ήρθατε. Δεν είναι η τελευταία φορά που βρισκόμαστε, δίχως άλλο. Σας ευχόμαστε καλή τύχη και αντοχή. Αντοχή, ναι. Σας ευχαριστώ κι εγώ. Λέει ο κύριος Κρεμονίνη. Πρόεδρος, ωραία. Διάφορα. Δεν έχουμε τίποτα. Οπότε έληξε η συνεδρίαση για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Α, η επόμενη συνεδρίαση θα λάβει χώρα στις 22 Μαρτίου, 9 με 12.30 και 3 με 6.30.